Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε παρακαλώ με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την έγκριση της δηλαδή. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη ως έχει. Σημείο 2. Έχουμε διερμηνία σήμερα από και προς 20 γλώσσες και μάλιστα έχουμε στείλει και το τα έγγραφα της συνεδρίασης ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-meeting και θα αναμεταδίδεται η συνεδρίασή μας και από το διαδίκτυο. Σημείο 3 της ημερής διάταξης. Να σας ενημερώσω ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015, 21 22 Δεκεμβρίου 2015 και 14 Ιανουαρίου 2016 ε, είναι έτοιμα προς έγκριση. Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσει μέχρι το τέλο της θα θεωρηθούν ω εγκεκριμένα. Για το σημείο 4 τώρα. Ε, ενημέρωση της Επιτροπής για την έκβαση των διοργανικών διαπραγματεύσεων για τα εξή ζητήματα. Το πρώτο θέμα αφορά τους ελέγχους και τις δραστηριότητες για την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών και τα μέτρα φυτοπροστασίας. Μέχρι ε, έχουμε την ευκαιρία στα τρία θεσμικά όργανα να υποβάλουν τις θέσεις τους σε σχέση με τα άρθρα για την χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων και να συζητήσουν τα πολιτικά, θέματα, τα πολιτικά ζητήματα του ελέγχου για τις εισρωές άρθρα 45 μέχρι 75, ε, για τα, τους ελέγχους της εισαγωγής, συγγνώμη. Έγιναν συζητήσεις σε επικοδομητικό πνεύμα και κρίθηκε ότι θα βρεθούν συμβαστικές τροπολογίες για τα περισσότερα θέματα. Μάλιστα για τα εκρεμή πολιτικά ζητήματα, το θέμα εκχώρησης εξουσιών θα ε, εξεταστεί σε ευρύτερο πλαίσιο. Δεύτερο θέμα, μείωση των εθνικών εκπομπών συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών ρήπων. Κατά τον πρώτο άτυπο τριμερή διάλογο της ε, οδηγίας για τα ανώτατα εθνικά όρια που έγινε στι 25 Φεβρουαρίου του 2016, το Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προέβησαν σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά πολιτικά θέματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2. Ε, ελαστικά πραγματικότητα, μεθάνιο και τον ενδιάμεσο στόχο για το 2025. Δεύτερος διάλογος, ε, τριμερής, έχει προγραμματιστεί για τις 4 Απριλίου 2016. Πέμπτο σημείο τη ημερήσης διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων της ε, Διατλαντικής Συμφωνίας ε, Εταιρική Σχέσης, το TTIP. Θα δώσω το λόγο στον αναπληρωτή διαπραγματευτή, τον κύριο Χίντο Χόμπεν. Του δίνω ένα δεκάλεπτο για την πρώτη του παρουσίαση. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Παρακαλώ κύριε Χόμπεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και καλημέρα σας. Ζητώ συγγνώμη γιατί ο επικεφαλής, το αφεντικό μου δηλαδή, ο κύριος Ιγνάσιο Μπερσέρο, απουσιάζει. Θα ζητά συγγνώμη γι' αυτό, θα κάνω ό,τι μπορώ να τον αντικαταστήσω επάξια. Νομίζω ότι τελευταία φορά που είχατε συζήτηση για την πορεία των διαπραγματεύσεων στη Συμφωνία TTIP ε, ήταν το Νοέμβριο. Οπότε θα ήθελα σήμερα να σας ενημερώσω για την πρόοδο που έχουμε πραγματοποιήσει έκτοτε και τις προοπτικές ε, για τους επόμενους μήνες του 2016 μέχρι το τέλος της ε, θητείας του Πρόεδρου Ομπάμα. Ως στόχο είχαμε θέσει ε, από το φθινόπωρο και για φέτος είναι κυρίως ο στόχος να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να καλύπτει όλα τα θέματα που είναι προς διαπραγμάτευση στο TTIP με στόχο να καταλήξουμε σε μια όριμη φάση των διαπραγματεύσεων μέχρι το καλοκαίρι. Προσπαθούμε να δρομολογήσουμε αυτή την προσπάθεια επιταχύνοντας το ρυθμό των διαπραγματευτικών γύρων. Είχαμε ένα γύρο τον Οκτώβριο, ένα το Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες, ένας θα γίνει τον Απρίλιο και ένας τέταρτος τον Ιούλιο. Σε κάθε τέτοιο διαπραγματευτικό γύρο προσπαθούμε να υποβάλουμε πακέτα προτάσεων και εμείς και οι Αμερικανοί που στη συνέχεια θα συνδυαστούν για να γίνουν συμβατές και να, να καταλήξουμε σε ενοποιημένα κείμενα. Αυτή η διαδικασία της ενοποίησης των κειμένων ε, ξεκινά με δύο ξεχωριστά κείμενα που μετά συνδυάζονται, γίνεται μια συμπίληση με στόχο να μειωθούν ε, οι εκκρεμότητες τα θέματα που βρίσκονται σε αγκύλες και με ένα συνεπή και συνεκτικό τρόπο ώστε να φτάσουμε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων, το end game που λέμε, με το μικρότερο δυνατό αριθμό πολιτικών κρεμοτήτων που θα εξεταστούν σε επίπεδο υπουργών. Από τον Νοέμβριο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ε, πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο σε δύο θέματα και στο νομοθετικό σκέλος και στο σκέλος των κανόνων. Ε, τρία είναι οι άξονε των διαπραγματεύσεων. Οι στι αγορές, ε, κανονιστική συνεργασία και συμβατότητα με τους κανόνες. Ε, έχουμε φυσικά πολλά κείμενα και το σχέδιο της σύμβασης που θα γίνει η συμφωνία TTIP που όπως θα φαντάζεστε θα είναι πολυσέλιδη, μπορεί να φτάσει μέχρι και τις χίλιες σελίδες, θα επιμερίζεται σε κεφάλαια και χάρη ενημέρωσης, θα έλεγα ότι η πιο σημαντική πρόοδος που πραγματοποιήσαμε από τον Νοέμβριο αφορά το νομοθετικό σκέλος, το κανονιστικό σκέλος, συγγνώμη, ε, που αφορά νέα κεφάλαια κανονιστικής συνεργασίας ε, και κανονιστικών πρακτικών και σε ό,τι αφορά ε, τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο, TBTs. Υπάρχουν κείμενα που είναι προσιτά και τα έχουμε στείλει και στο Κοινοβούλιο και σε αυτά προσπαθούμε να λάβουμε στο έπακρο υπόψη τους, τους στόχους και τις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στο ψήφισμα του, του Ιουλίου, της 8 Ιουλίου του 2015 για το TTIP και επίσης να λάβουμε υπόψη και τις συστάσεις των ε, επιμέρους κοινοβουλευτικών επιτροπών και της δικής σας φυσικά που κατέληξαν στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το TTIP. Από τον Νοέμβριο επίσης υποβάλαμε και ένα κείμενο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αηφόρο ανάπτυξη. Τις δεσμεύσεις δηλαδή στα θέματα απασχόλησης και περιβάλλοντος όπως λένε οι Αμερικανοί. Το περιμέναμε πώς και πώς αυτό το κείμενο και ήταν ένα είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα των διαπραγματεύσεων στο μέτρο που θέλουμε μέσω των δεσμεύσεων για την εργασία και το περιβάλλον να δείξουμε ότι και οι Ηνωμένε και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να ασκήσουν ή να έχουν ένα κοινό όραμα ε, ηγετικού ρόλου ώστε να προωθήσουν παγκοσμίω ένα υψηλό επίπεδο δεσμεύσεων για την εργασία και το περιβάλλον. Σχεδόν πρωτόγνωρο για τέτοιου είδους εμπορική συμφωνία. Υπάρχει λοιπόν μια ποιοτική πρόοδος, ένα ποιοτικό άλμα. Θα το διαπιστώσετε αυτό διαβάζοντας το κείμενο για την αηφόρο ανάπτυξη και μάλιστα τρεις μήνες μετά το γύρο των Βρυξελών απάντησαν οι Αμερικανοί με ένα δικό τους κείμενο σε σχέση με το δικό μας και προσπαθούμε τώρα να ενοποιήσουμε αυτά τα δύο κείμενα. Τώρα, τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Υπάρχουν ακόμη κάποιοι τομείς με εκκρεμότητες. Γι' αυτούς θα πρέπει και οι δύο πλευρές να συνεχίσουν μέχρι το καλοκαίρι τις διαπραγματεύσεις για να αναπτύξουν σχέδια κεφαλαίων ή σχέδια παραρτημάτων. Και νομίζω από τους πιο σημαντικούς τομείς αφορά το συγκεκριμένο έργο ανακλάδο, ανατομέα, στο κανονιστικό σκέλος. Και όταν μιλώ για τομείς εννοώ εννέα τέτοιους κλάδους. Ε, προδιαγραφές ασφάλειας για τα οχήματα είναι ένας ας πούμε. Ή ε, επιθεωρήσεις και έλεγχοι για φαρμακοβιομηχανίες, καλλιτικά, χημικά, παραστοκτόνα και μια σειρά τέτοιων τομέων για τους οποίους έχουμε θεσπίσει κάποιους στόχους για τους επόμενους μήνες. Και κατά την εκπόνηση των στόχων αυτών προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη πλήρως το κανονιστικό πλαίσιο του κάθε κλάδου που μερικές φορές είναι πολύ διαφορετική μεταξύ τους, όπως τα χημικά για παράδειγμα. Και προσπαθούμε έτσι να βελτιώσουμε την ποιότητα των μελλοντικών νομοθετικών διατάξεων, χωρίς όμως να επηρεάζουμε είτε την ε, κανονιστική αυτονομία η κυριαρχία είτε τις ε, το, ε, εθνικές διατάξεις ή σε καμία περίπτωση να μην υποβιβάσουμε τις υψηλές προδιαγραφές και πρότυπα προστασίας. Το τονίσαμε αυτό και το διατρανώσαμε και στο Κοινοβούλιο και προς την κοινή γνώμη, διευκρινίζοντας τους στόχους μας για το TTIP σε τομείς που ίσως υπάρχουν διαφορές στην νομοθεσία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, να επιστήσω την προσοχή σας στην επικείμενη δημοσίευση της ενδιάμεσης ε, μελέτης βιωσιμότητας για το TTIP. Την έχει ολοκληρώσει μία Ολλανδική εταιρεία συμβούλων με έδρα το Ελπίζουμε το πρώτο σχέδιο να ολοκληρωθεί σύντομα και να δημοσιευθεί τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για μια ενδιάμεση τέτοια μελέτη βιωσιμότητας του TTIP. Θα υποβληθεί σε έλεγχο και θα οριστικοποιηθεί προς τα τέλη του έτους και θα εκτιμά τον αντίκτυπο μιας πιθανής συμφωνίας στη ΤΥΠ σε όλους τους τομείς της οικονομίας στα κράτη-μέλη. Και ένα τελευταίο σχόλιο για το πού βρισκόμαστε τώρα στην διαπραγματευτική διαδικασία. Έχουν περάσει δυόμιση χρόνια από την έναρξη των διαπραγματεύσεων και προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τις διαπραγματεύσεις ε, ως διαπραγματεύσεις με αρχή, μέση και τέλος. Το τέλος, τελική φάση, το endgame, θα ασχοληθεί με τα πιο ακαθόδη και ευαίσθητα ζητήματα. Τώρα βρισκόμαστε στο middle game, αυτό που λέμε, στη μεσαία φάση των διαπραγματεύσεων. Προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε όσο ε, περισσότερες δεσμεύσεις για πρόσβαση στις αγορές και για να έχουμε μια αποτελεσματική τελική φάση των διαπραγματεύσεων με όσο το δυνατό μικρότερο αριθμό εκκρεμών θεμάτων. Φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε μια τελική φάση των διαπραγματεύσεων ε, ανοιχτή προς όλες τις κατευθύνσεις με πληθώρα εκκρεμών θεμάτων. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει η προεργασία και η διεκπαιρέωση ως το δυνατόν περισσότερο θεμάτων σε προηγούμενη φάση, την ενδιάμεση φάση των διαπραγματεύσεων. Γιατί ε, στο μεταξύ θα έχουμε αναπτύξει κείμενα εκεί που δεν υπήρχαν, θα ενοποιήσουμε προτάσεις μεταξύ των δύο εταίρων στις εκκρεμότητες και θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον αριθμό των ε, αγγελών ε, ώστε να καταλήξουμε σε μικρό αριθμό θεμάτων για την τελική φάση. Πάντως πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε σημαντικό αριθμό κεφαλαίων πριν περάσουμε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων, στο endgame. Επίσης και εμείς και οι Αμερικανοί εταίροι ε, είμαστε προσιλωμένοι στη διατήρηση αυτής της ε, όθης που έχουμε δώσει στη διαδικασία και στο γοργό ρυθμό. Είναι άλλωστε η τελευταία χρονιά της ηττίας Ομπάμα. Ε, θα βρίσκεται στην εξουσία μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 2017. Ο Μαρκ Φρόμαν, που είναι ο επικεφαλής των ΗΠΑ στη έχει και δημοσίως αναλάβει την υποχρέωση να προσπαθήσει να διεκπαιρεώσει φέτος στις διαπραγματεύσεις για το TTIP, ε, όσο είναι στη θέση του δηλαδή, και εμείς ε, έχουμε δεσμευτεί να παρακολουθήσουμε αυτό το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που θα θέσουν οι Αμερικανοί, υπό την επιφύλαξη βέβαια ότι θα φροντίσουμε η ουσία να ε, επικρατεί της διαδικασίας. Δεν πρόκειται δηλαδή να επισπεύσουμε τις διαπραγματεύσεις εις βάρος της ποιότητας των δεσμεύσεων, εις βάρος της ουσίας. Γιατί η ουσία προέχει για μας. Και η ποιότητα προέχει και προηγείται της ταχύτητας. Πάντως, υπό την επιφύλαξη εξασφάλισης ποιότητας και της ουσίας, είμαστε κι εμείς ε, προσιλωμένοι στο στόχο της επίτευξης της σταθερής πρόοδου. Έχουμε πολύ δημόσιο έλεγχο ε, και τεράστιες ε, πολιτικές επενδύσεις στην Ευρώπη στα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από, τις ευρωπαϊκ... από και θέλουμε και εμείς να υποβάλουμε στο δυνατό περισσότερα κείμενα και να, προλιάνουμε, να λιάνουμε τις διαφορές με τους Αμερικανούς. Πάντως, τους τελευταίους μήνες έγινε εντυπωσιακή πρόοδος και θα διαπιστώσετε τους σε πολλούς τομείς που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και τη δική σας επιτροπή, κυρίως όμως τα κεφάλαια για τις δεσμεύσεις, για την εργασία και το περιβάλλον, το κεφάλαιο δηλαδή της αηφόρου ανάπτυξης, εκεί είναι που σημειώσαμε την πιο εντυπωσιακή πρόοδο από τον Νοέμβριο. Γιατί τώρα έχουμε περάσει σε συγκεκριμένα κείμενα στο ευρύτερο αυτό κεφάλαιο και μπορείτε να τα εξετάσετε και να δείτε σε ποιο βαθμό οι παράμετροι και οι συστάσεις που μας δώσατε τους τελευταίους μήνες συμπεριλήφθησαν στην ευρωπαϊκή πρόταση. Νομίζω ότι από αυτήν την άποψη επιτελέσαμε καλά το έργο μας. Θα, θα το κρίνετε όμως εσείς. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε συνεδρίες και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τον γύρο των έρωτα απαντήσεων. Να δώσουμε το λόγο καταρχά στον κύριο Ντόρφμαν, ο οποίο είναι ο μόνιμο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε. Σα ευχαριστούμε για τι πληροφορίε αυτέ. Είναι νομίζω πολύ ωφέλιμε και σίγουρα στην Επιτροπή μα ε, τι χρειαζόμαστε τέτοιε ενημερώσει ε, τακτικά. Ε, μία ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα. Το θέσατε και εσεί το θέμα, αγαπητή κυρία. Σε ποιο βαθμό βλέπετε στις διαπραγματεύσεις ε, ε, τον αντίκτυπο της προεκλογικής εκστρατείας στην Αμερική. Πώς ε, λοιπόν επηρεάζει αυτή η κατάσταση τις διαπραγματεύσεις για το TTIP και οι δύο υποψήφοι, οι δύο μεγάλων κομμάτων στη ΣΥΠΑ. Ναι, λίγο πολύ πλέον ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Και δήλωσαν και δύο εξίσου πρόθυμοι να προωθήσουν το TTIP. Επηρεάζει λοιπόν αυτό τις διαπραγματεύσεις. Ποια είναι η άποψή σας. Τούτου λεχθέντο, Να υπογραμμίσω εκ νέου τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, την οποία και καταρτήσαμε πριν από κάποιες εβδομάδες για το TTIP και εδώ θα ήθελα να, να επισημάνω τρεις τομείς. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ρυθμιστική συνεργασία ρυθμιστική συνεργασία η οποία θα μπορούσε λογικά να οδηγήσει σε εξίσωση προς τα κάτω ή προς τα πάνω των προτύπων. Σε πολλούς τομείς από ευρωπαϊκής πλευράς έχουμε συμφέρον να εξισωθούν προς τα πάνω. Στο δικό μας επίπεδο τα πρότυπα, οι προδιαγραφές αυτές γιατί πολλοί από αυτούς τους τομείς μας απασχολούν ιδιαίτερα, όπως για παράδειγμα τα θέματα ασφάλειας τροφίμων. Εδώ σαφώς έχουμε πιο υψηλά πρότυπα από ό,τι της είπα. και αν θα υπάρχει μεγαλύτερη ρυθμιστική συνεργασία θα πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση ότι θα προσαρμοστούμε στα δικά μας πρότυπα. Δεύτερη ερώτηση για την φυτοπροστασία. Δεν επαναφέρατε το θέμα. Σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των τροφίμων υπάρχουν διάφορες, ε, διάφοροι περιορισμοί. Αλλά εδώ μιλάμε πιο πολύ για προδιαγραφές ε, και νομοθεσία για την φυτοπροστασία. Τι γίνεται λοιπόν εδώ. Υπάρχουν υποχωρήσεις και από αμερικανικής πλευράς, όπου ισχύουν ε, κάπου και παράλογες ρυθμίσεις, για παράδειγμα μηδενική ανοχή και σε ό,τι αφορά μια μεγάλη σειρά τέτοιων μέτρων φυτοπροστασίας, εμπορικές, ε, εμπορικοί περιορισμοί. που θα πρέπει να περιοριστούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, αν θέλουμε να υπάρχουν εξαγωγές τροφίμων από την Ευρώπη προς τις είπα Τρίτο, τρίτο θέμα, η προστασία του καταναλωτή και η ασφάλεια των τροφίμων. Σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια των τροφίμων, θέλουμε να στηριχθούν τα δικά μας ε, πρότυπα σε ό,τι αφορά την πλανοποίηση, τη χρήση ορμόνων, σε ό,τι αφορά το βόλιο κρέας κτλ. Σίγουρα θα θελήσουμε μια σχετική ρύθμιση. Σίγουρα θα θέλουμε απαγόρευση εισαγωγών τέτοιου κρέατος που έχει περάσει ορμονοθεραπεία. Τελικό θέμα, η χημική επεξεργασία και τα σχετικά πρότυπα. Είπαμε στην γνωμοδότησή μας ότι δεν θέλουμε να υπάρχει εξίσωση προς τα κάτω ή να θέσουμε ένα αμφιβόλο το REACH. Τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις αυτές, ποια είναι η αντίδραση των ΗΠΑ τουλάχιστον πώς αντιδράει η διαπραγματευτική ομάδα τον είπα, για το θέμα αυτό. Αυτά ως προς τις ερωτήσει μου. Θα ήθελα επί της, αρχή να, επί της αρχής να διευκρινίσω το εξή. Πάντα υποστηρίζα ότι αν ε, πετύχουμε μία συμφωνία η οποία θα έχει θετικό αντικτύπο στο εμπόριό όμως αυτό είναι πολύ θετικό αλλά να μην αφήσουμε την κυβέρνηση Ομπάμα να μας πιέσει, επειδή έχει μόνο λίγους μήνες στη διάθεσή της ακόμα, να τα πασαλείψουμε όλα αυτά. Η εξαγωγή τροφίμων, για παράδειγμα, πέρσι από Ευρωπαϊκή Ένωση προς ΕΠΑ πήγε πάρα πολύ καλά, σημειώθηκε σημαντική και καλή αύξηση δεν ε, μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι χάνουμε σε ό,τι αφορά το εμπόριο με τη ΣΥΠΑ. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εμείς είμαστε οι πιο ωφελούμενοι, αλλά φυσικά μπορεί να βελτιωθεί και περαιτέρω η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν να ε, μην αφήσουμε να μας πιέσουν οι πολιτικές συνθήκες της ΣΥΠΑ και ο Πρόεδρος ο και να πετύχουμε μια κατάσταση win-win. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπάλας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, Επιτροπή μας και την, ε, την Ευρωπαϊκή Μάλλον Επιτροπή και τον εισηγητή μας για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Καταρχάς να εκφράσω τη συμφωνία μου με τον εισηγητή σε αυτό το στάδιο για το γεγονός ότι για τα θέματα του TTIP πρέπει να δούμε κατά πόσο η συμφωνία αυτή ε, έχει να κάνει με τα συμφέροντά μας ή όχι. Οι σχέσει μα αυτή τη στιγμή με τι ΗΠΑ και οι δραστηριότητε των ΗΠΑ πρέπει να είναι καταστροφικέ από πλευρά ε, παγκόσμια κλίμακα. Πρέπει λοιπόν να δούμε την όλη κατάσταση. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάτι που υπόθηκε ιδίω για την ε, ανακοίνωσή του στην εξαγγελία του ότι θα γίνει μελέτη αντικτύπου. Ήθελα να μου πούν ακριβώ ποιοι θα είναι οι στόχοι αυτή τη μελέτη αντικτύπου. Να εξετάσουν το σύνολο των πεδίων διαπραγμάτευση, μελέτη αντικτύπου που θα εντοπιστεί σε πιο συγκεκριμένα θέματα με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια ή τέλο πάντων θα έχει κάποια συγκεκριμένα σημεία στα οποία θα επικεντρωθεί. Ήθελε επίση να ξέρω αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ποιο θα την εκπονήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει να μπορέσουν και εμπειρογνώμονες από διαφορετική προέλευση να συνεργαστούν στον συλλογικό σκοπό ή θα είναι απλώς ε, άνθρωποι που συμμετέχουν ήδη στις διαπραγματεύσεις και που θα εμπλακούν στην ε, σύνταξη αυτής της μελέτης. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να έχουμε την καλύτερη δυνατή παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστούμε κυρία Μιούλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτά που μας ε, είπατε. Ξέρω ότι υπάρχει ένα ευρύ κίνημα στη Γερμανία κατά του TTIP και καθημερινά προστίθενται άτομα σε αυτό το κίνημα και φυσικά ανακύπτει και το ερώτημα όπως και το είπε και ο κύριος Ντόρφμαν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τι γίνεται με τους συνηθικά τροποποιημένους οργανισμούς, τι γίνεται με τις ορμόνες, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι εισαγωγές τροφίμων από τη ΣΥΠΑ ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια συζητήσαμε τη νέα νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Τι γίνεται με τη χρήση αντιβιωτικών στην εκτροφή ζώων στις ΙΠΑ. Ε, Μπορούμε εδώ να ασκήσουμε επιπλέον ε, μάλλον θα μπορούσε να προκύψει τελικά επιπλέον πίεση για τους Ευρωπαίους εκτροφείς. Και είναι σημαντικό επειδή υπάρχει και ένα έγγραφο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της, της παράνομης υλοτομίας. Πώς αξιολογείται την Ευρωπαϊκή Δασοκομεία και τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι στα πλαίσια των τρέχουσων διαπραγματεύσεων δεν θα προκύψει σίγουρα πίεση στους Ευρωπαίους εκτροφείς λόγω των διαφορετικών προτύπων ως προς την εκτροφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριο Στάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θυμάμαι που ήμουν εισηγητής ε, στο ψήφισμα του Ιουλίου που ψηφίσαμε πέρσι τον Ιούλιο. Και θυμάμαι τότε στη συζήτηση που Είχαμε και ακούσαμε το Δεκέμβριο του 2014 μία ομιλία της κυρίας Μάλμστρομ η οποία το είπε τότε και το επανέλαβε και μετά με σαφήνεια ότι με τι είπα υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικά επίπεδα ε, νομοθεσίας σε διάφορους τομείς και ότι αυτή η διαφορά ποιότητας είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορέσει ποτέ να πετύχουμε συμφωνία. Το TTIP μιλάει για τις μη δασμολογικούς ε, φραγμούς. Αλλά αυτά είναι τα δικά μας θέματα, τα πράγματα που αποφασίσαμε με δημοκρατικό τρόπο εδώ στο Κοινοβούλιο, για τα οποία πολεμήσαμε, τα διαπραγματευτήκαμε με τα Υπουργικά Συμβούλια και με πολύ δημοκρατικό τρόπο λοιπόν προέκυψαν αυτοί οι μη δασμολογικοί φραγμοί. Μας λέει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας το λέει και σε κάθε συνάντηση και συζήτηση ότι μιλώντας με τους Αμερικανούς για τους μη δασμολογικούς φραγμούς ε, δεν πρόκειται να περιορίσουμε τα δικά μας πρότυπα. Μα στην πραγματικότητα, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήδη τώρα σε μια σειρά τομέων ρίχνουμε τα πρότυπά μας. Και έχω υπόψη μου τη συζήτησή μας για τους παθογόνους οργανισμούς στο κρέας. Έχω υπόψη μου τη συζήτησή μας ε, για την κλωνοποίηση. Μας είπε ο κύριος Λίζε ότι μετά από τις διαπραγματεύσεις για το TTIP οι απαιτήσει από πλευρά της Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που θα θέλαν. Πολύ. τι γίνεται με τον κανονισμό για την καθαρή βενζίνη, το όλο πακέτο για το Better Regulation. Όλα αυτά είναι μέλος του, μέρος του Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα πρότυπά μας, να μην τα ρίξουμε στο ψήφισμα του Ιουλίου του 2015 το Κοινοβούλιο με μεγάλη σαφήνεια διακήρυξε ότι δεν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί για κάποιου τομεί σε ό,τι αφορά του γενετικά τραποποιημένου οργανισμού, σε ό,τι αφορά τι ορμόνε, την κλωνοποίηση, το REACH. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά το REACH, αλλά και την εφαρμογή του REACH. Και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για το REACH. Εγώ να πιστέψω ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων δεν θα επηρεάσει το REACH, αλλά το θέμα είναι και η εφαρμογή του REACH. Γιατί βλέπουμε σήμερα ήδη ότι ο κόσμος πηγαίνει στο Ελσίνκι για να διαπραγματευτεί θέματα εφαρμογή. Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα είναι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας το εγγυηθεί, γιατί ξέρουμε ότι είναι αντικείμενο αυτό διαπραγματεύση. υπάρχουν διαρροές. Μπορεί να μας πει λοιπόν με αφήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον υπάρχει διαπραγμάτευση για την εφαρμογή του ναι ή όχι, και τι μπορούμε να περιμένουμε. Τελευταίο ζήτημα, μια μεγάλη διαμάχη στο Κοινοβούλιο ήταν η συζήτηση για το ISDS. Investment States Dispute Settlement για το σύστημα α, συλλογικών αγωγών. Ξέρουμε ε, ότι υπάρχει και μια πρόταση της κυρίας Μάλμστρομ επιτάπητος προς διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Ας μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν που βρισκόμαστε, πώς αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί την πρόταση, είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Γιατί φυσικά το ζήτημα που εξακολουθεί να είναι εκρεμές είναι το εξή Το IS είναι μια διακοσμητική αλλαγή σε σχέση με το ISDS. Το θέμα είναι ότι οι αλλοδαποί επενδυτές θα έχουν πιο πολλά δικαιώματα από τους εμεδαπούς. Είναι δυνατόν να το εγκρίνει αυτό το κοινοβουλίο μας. Εμείς είμαστε ξεκάθαρα αρνητικοί. Thank you very much, Mr. Balzo. Elnök úr, köszönöm a szót. Nyilván ennek a nem az a... κύριος Μπάλτσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σκοπός ε, του θέματος αυτού στην ημερήσια διάταξη δεν ε, είναι να σας αναλύσω γιατί πιστεύω ότι θα την αρνητική σύναψη μιας συμφωνίας μπορούμε να σκεφτούμε και πόσο φιλόδοξος θα μπορούσε να είναι ο πρόεδρος Ομπάμα στην ε, όλη εκστρατεία και διακηρύσει ότι θέλει να ολοκληρωθεί η σύναψη της συμφωνίας και ότι θα ωφεληθούν και οι αμερικανικές εταιρείε. Δύο ερωτήσεις λοιπόν έχω. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ε, δικαστικών επιλύσεων. Η πρόταση κατά την οποία δεν έγινε δεκτή η λύση του ISDS απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο. Υπήρξε μια άλλη πρόταση λοιπόν που συμπεριλάμβανε διάφορα στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση του το ICDS για τα επενδυτικά δικαστήρια. Κατά δεύτερον, το 2014 απευθύνθηκε από τα Εθνικά Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 20 Εθνικά Κοινοβούλια, μια ερώτηση προς το, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν τα κράτη-μέλη θα υποχρεωθούν να επικυρώσουν την ε, συμφωνία αυτή. Η συνθήκη της Λισαβόνας λοιπόν προβλέπει νομική ο ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία δεν θα έπρεπε και δεν θα υποχρεούντουσαν τα εθνικά κοινοβούλια να επικυρώσουν ή θα μπορούσε να ισχύει μια μεικτή ε, ένα μεικτό σύστημα επικύρωσης. Ε, τι θα ισχύσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτές τις δύο ερωτήσεις λοιπόν έχω να κάνω. Το θέμα του ISDS για τις ε, την επίλυση διαφορών κράτους επενδυτή και για το θέμα της μεικτής ή μη επικύρωσης. Τώρα, να σας πω ότι είμαι μη εγγεγραμμένος και πρέπει να πω ότι με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω ότι ποτέ δεν έχουν απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ερωτήματα που του απευθύνω. Κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενημέρωση που μας έκανε για την ε, πορεία των διαπραγματεύσεων, τον κύριο Χόουμπεν. Μας ε, παρουσίασε αρκετά νέα στοιχεία και χαίρομαι που έλαβε υπόψη και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το TTIP με τις θέσεις μας. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως είδαμε και από τις πρόσφατες εκλογές στη Γερμανία, οι Ευρωπαίοι πολίτες λοιπόν εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι ασύμετρο αυτό το μοντέλο σχέσεων και άνισο. Θα πρέπει λοιπόν να δισκεδάσουμε τις αφιβολίες και τις ανησυχίες των συμπολιτών μας. Βέβαια σε υψηλό πολιτικό επίπεδο μας διαβεβαιώνεται και μας καθησυχάζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υποβιβαστούν οι προδιαγραφές μας, οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές στην διαπραγματευτική διαδικασία. Χρειαζόμαστε όμως και μια νομική βάση για να ε, αποτρέψουμε μια τέτοια υποβάθμιση. Στις αρχές του έτους, ή μάλλον πέρυσι, επισκεφθήκαμε με συναδέλφους ε, της Ηνωμένε Πολιτείε και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων ε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε πάρα πολλά θέματα και οι ευαισθησίες μας είναι διαφορετικές. Για την κλωνοποίηση, τι χημικές ουσίες, ε, του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμούς υπάρχει μεγάλο χάσμα απόψεων μεταξύ μας. Επίσης έχουμε από τη μια τις Ηνωμένες που είναι μια συμπαγής ε, οντότητα και την, από την άλλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ένωση 28 διαφορετικών ε, χωρών μελών και μάλιστα πολλές έχουν ε, πολλές επιφυλάξεις για τις αντιλήψεις των Αμερικανών, για τα μεταλλαγμένα, για την κλωνοποίηση και το καθεξής. Νομίζω ότι υποτιμούμε τη σοβαρότητα αυτών των διαφορών. Αν κατάλαβα καλά, η αμερικανική πρόταση προβλέπει και οι περιβαλλοντικοί κανόνες να υπόκειται στον μηχανισμό ISDS, δηλαδή της επίλυσης διαφορών κράτους επενδυτή. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτό το αμερικανικό αίτημα. Πώς ε, πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαφυλάξει τις περιβαλλοντικές μας προδιαγραφές σε περίπτωση διαφοράς με τους Αμερικανούς. Επίσης, ε, μιλήσατε για κανονιστική αυτονομία. Πώς ε, θα μπορέσουμε παρά τους νέους μηχανισμούς του ISDS να προασπίσουμε αυτή την ε, κανονιστική μας αυτονομία και να μπορούμε και στο μέλλον ακόμη και να αναβαθμίσουμε τις προδιαγραφές και τα πρότυπά μας. Θα ληφθεί δε όντως υπόψη η περιβαλλοντική ευαισθησία των κρατών μελών. Αυτά ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε, κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το παρακολούθησα, το, το θέμα αυτό πολύ στενά και με την συνεργασία με τον κύριο Στάς και παρακολουθώ λοιπόν πάρα πολύ, καλή, πολύ, πολύ καλά τις ε, διαπραγματεύσεις. Και μελετώ πάρα πολύ τα πράγματα, τα έγγραφα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να είναι τόσο εμπιστευτικά και απόλυτα. Διαπιστώνω λοιπόν ότι, ότι αυτά που είπε ο κύριος Πέτερλε μόλις, αυτά που βλέπουμε ως τώρα πιστοποιούν ότι είναι ασύμετρες οι διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει, ορίζει κάποιες θέσεις και οι ΙΠΑ εμένουν στη θέση του, στην αρχική. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Είναι λοιπόν εντελώς ασύμετρες οι διαπραγματεύσεις, όπως και το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε πετύχει έως τώρα. Δεν μπορούμε να πείσουμε για κάτι διαφορετικό την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Και σε κάποιους τομείς βλέπουμε ότι σήμερα δεν είναι δυνατόν να πετύχουμε συμφωνία ήδη σήμερα. Το παραδέχεται αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ απλά δεν είναι δυνατόν να πετύχουμε συμφωνία χωρίς να αλλάξουμε την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει η νομοθεσία, αλλά πολύ φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περάσει και θα αλλάξει κάποια βήματα σε ό,τι αφορά τους εφαρμοστικούς κανονισμούς. Αλλά έχουμε και δημοκρατικό έλεγχο και δεν μπορώ να καταλάβω πώς σήμερα ε, ε, επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυτοπροστατευτικά τα οποία δεν θα έπρεπε να επιτρέπει. Πώς ε, μπορεί να επιτρέψει, για παράδειγμα, στοιχεία σε, στα τρόφιμα τα οποία επίσης δεν έπρεπε να επιτρέπονται. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν μια πολύ προσεκτική ανάλυση και αν κάνουμε την ανάλυση αυτή θα καταλάβουμε ότι μας ε, έχουν στριμώξει για να προσαρμοστούμε στα δικά τους πρότυπα. Παρά όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση γιατί είναι πραγματικά πολύ αρνητικό. Ένα άλλο πόρισμα της ε, επισκεψής μας. Ένας άλλος τομέας όπου δεν έχει αλλάξει επίσης ε, τίποτα είναι ο εξής. Οι είπα δεν μπορούν να μας εγγυηθούν ότι υποχρεούνται να εγγυηθούν αυτά που θα συμφωνήσουμε στις διαπραγματεύσεις να εφαρμοστούν σε υποομοσπονδιακό επίπεδο. Δηλαδή αυτά που συμφωνούμε δεν μπορεί να δεσμευτεί η ομοσπονδιακή οι ομοσπονδιακές αρχές ότι θα εφαρμοστούν σε επίπεδο πολιτιών. Τι νόημα έχει λοιπόν να κάνουμε διαπραγματεύσεις για το TTIP αν οι μεμονωμένες πολιτείες δεν δεσμεύονται πολύ απλά. Αλλά ας μην είμαστε μόνο αρνητικοί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τουλάχιστον σε κάποιους τομείς επιτέλους κατάφεραν να αντισταθούν στην ε, βορειοαμερικανική νοοτροπία. Σε ό,τι αφορά τους διαταράκτες, για παράδειγμα. όπου ασκούταν εμπορική πίεση. Και πραγματικά βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανθίσταται. Το παρατηρώ αυτό, τα παρακολουθώ όλα αυτά τα νομοθετικά και νομίζω ότι εδώ δείχνει μια θετική πτυχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ασύμετρος χαρακτήρας στις διαπραγματεύσεις. Και αυτό σίγουρα θα μας προβληματίσει και στο μέλλον και το θέμα το ότι η ομόσπονδη κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να δεσμευστεί για τα πολιτείε θα μας απασχολήσει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκέρινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς να κάνω μια δήλωση τρόπον ότι με ενδιαφέρει πολύ να, να επιτύχουμε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις TTIP Νομίζω ότι οι εμπορικές μας σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι ζωτική σημασία για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Και για μένα ως Βρετανή ε, βουλευτή είναι ένα θέμα που είναι καυτό εν ώψη του δημοψηφίσματος για την παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το θέμα είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας δώσει πρόσβαση σε αγορέ εξαγωγών. Με ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ να επιτύχουμε μια καλή συμφωνία στο δυνατόν συντομότερο. Και το λέω ε, αυτό ευθύς εξ αρχής για να εξαγγείλω ε, τα όσα έχω να πω με μεγαλύτερη ευκολία. Διότι ο στόχος μου δεν είναι καθόλου να μπλοκάρω τις συμφωνίες TTIP. Την διαπραγματεύσει μέλλον TTIP. Όμω, και επιμένω σε αυτό, θα πρέπει να έχουμε λεπτομέρειε για το πώ, ιδίω για το θέμα του, των πεδίων ε, που, και των τομέων ενδιαφέροντος που αφορούν την Επιτροπή μας, μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία συμβατεί με τα συμφέροντά μα. Διαρκώ ακούμε, και δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω ότι υπάρχει καλή πρόθεση πίσω από αυτό, ότι θα βεβαιωθούμε ότι τα πρότυπά μα δεν θα υποβαθμιστούν. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε φτάσει, πολύ, έχουμε σχεδόν φτάσει στο σημείο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επόμενη παρουσίασή τη για τη θα πρέπει να μα δώσει εξηγήσει για το ακριβώ ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί για να επιτύχουμε αυτήν την συμβατότητα με τα δικά μας τα πρότυπα την αντιστοιχία. Πραγματικά δεν αμφισβητώ την καλή πρόθεση, όμως πώς θα εκφραστεί αυτό. Και εφόσον βρεθεί τρόπο να εκφραστεί, θα πρέπει να δούμε αυτά τα κεφάλαια ξεχωριστά ενδεχομένω. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει την ευκαιρία να τα εξετάσει όλα αυτά. Οι απόψει μα θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Ιδάλω θα ήταν ε, πραγματικά τραγελαθικό αυτή η συμφωνία να εξαρτάται από την τοποθέτηση των κοινοβουλίων και να απορριφθεί, ενώ είχαμε την ευκαιρία να τα δούμε εκ των προτέρων. Όπω είπα λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μα δώσει λεπτομέρειε για να μα εξηγήσει ποιου ακριβώ μηχανισμού έχει ενεργοποιήσει. Ευχαριστούμε κυρία Γιατανάκη. Ευχαριστούμε πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή και τον Εισαγητή για τις πληροφορίες του, όμως θα χρειαστώ πολύ περισσότερα στοιχεία για να είμαι σε θέση να αξιολογήσω την κατάσταση ε, και το πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα. Δεν είμαι λοιπόν σε θέση να σας πω εάν τα πράγματα πάνε καλά ή όχι, έτσι όπως τα βλέπουμε. Μιλήσατε για την πτυχή της ρύθμισης και φαίνεται ότι έχετε κάνει πολλά βήματα πρόοδου. Τι θα πει όμως ρυθμιστική προσέγγιση. Ότι μπορείτε τα πρότυπα να τα αναβαθμίσετε μεν, αλλά μπορείτε τα, όποτε θέλετε και να τα υποβαθμίσετε. Μας ενδιαφέρει λοιπόν σε ποιες διατάξεις υπάρχει μια τάση να δούμε τα πρότυπά μας και να τα κάνουμε και καλύτερα, όπως με τα αντιβιωτικά ή τα τρόφιμα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται με την προστασία των καταναλωτών. Δεν μου αρκεί να μου λέει κανείς ότι θα μπορούσαμε ή να τα βελτιώσουμε ή να τα υποβαθμίσουμε τα πρότυπά μας. Τι ακριβώς κάνετε, αυτό μας ενδιαφέρει. Ακούμε ότι έχετε κάνει κάποια βήματα πρόοδο, αλλά ποια είναι αυτά. Ακριβώ δηλαδή τι συμβαίνει με την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών. Εκεί μα ενδιαφέρει ακριβώ να ξέρουμε τι βήματα συγκεκριμένα πρόοδο επιτύχατε και με ποιο τρόπο. Διαπραγματεύσει για τι τιμέ έγιναν ή καθόλου δεν το έχετε αγγίξει αυτό το θέμα. Τι ακριβώ έχει γίνει σε αυτό το τομέα. Τρίτη ερώτηση. Σε ποιου τομεί δεν υπήρξαν καθόλου βήματα πρόοδου. Ποια είναι τα ζητήματα που δεν ε, αγγίξατε καν. Ψεύρισκονται βρίσκονται σε ακριμότητα γιατί ακόμη υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλήσεις απόψεων. Άλλη ερώτηση και αυτή σημαντική. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μας ακολουθούν στην όλη μας διάθεση να αναβαθμίσουμε τα πράγματα. Είναι συνεργάσιμοι Διότι, όπω ξέρετε, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και την κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτείων. Και όπω έχουμε πει για την περίπτωση των διαπραγματεύσεων για άλλα σημεία, δεν σημαίνει ότι σε ομοσπονδιακό επίπεδο οι Πολιτείε και εκείνοι του γνώμη ακολούθησαν ε, τις... την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων TTIP. Η κυβέρνηση, λοιπόν, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ε, δεσμεύονται να λάβουν υπόψη την άποψη των πολιτών. Είναι αυτό κάτι που θα παίξει ρόλο ή όχι. Αυτές τις ερωτήσεις θέλω να σας θέσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Καρδίνη. Ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία και να θυμίσω αλλά φαίνεται και ακούγεται και από τις σημερινές παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο φαίνεται όλοι να συγκλίνουν προς το γεγονός ότι δεν θέλουμε οι διαπραγματεύσεις να γίνονται κρυφά. Το δείξαμε και στην περασμένη θητεία όταν ε, μπλοκάραμε την ε, ε, προηγούμενη συμφωνία για τη μορφή της, διότι δεν υπήρχε διάθεση να βρεθεί λύση για, τον, για το επεξεργασμένο κρέας. Εδώ λοιπόν οι μεγαλύτερες μας ανησυχίες επικεντρώνονται στα θέματα αρμοδιότητα τη επιτροπή μα, για την δημόσια υγεία, την επιστηστική ασφάλεια, την ε, καλή υγεία των ζώων και των φυτών και τι πληροφορίε προ τους καταναλωτέ. Είναι προφανές, το θύμισε και η συνάδελφο Γκίρλινγκ, ότι προφανώς ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτευχθεί αυτή η εμπορική συμφωνία. Όμως από την άλλη είναι εξίσου αληθές ότι το να είναι έγκυρη η συμφωνία και ουσιαστική μας ενδιαφέρει. Η αμερικανική προσέγγιση και η ευρωπαϊκή σίγουρα διαφέρουν ε, κατά πολύ. Σκεφτείτε την αρχή της προφύλαξης που εφαρμόζουμε στην Ευρώπη ή τους ελέγχους που, που διεξεγάγουμε. Εμείς έχουμε μια στρατηγική την οποία έχουμε συζητήσει επί μακρόν. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία εκμελασιμότητα. Οι Αμερικάνοι δεν κάνουν τα, μισά από αυτά. Επίσης δύο ζυζανοκτώνα τα οποία ζυζανιοκτώνα τα οποία στην Ευρώπη έχουν απαγορευτεί, όμω στι Ηνωμένε Πολιτείε επιτρέπονται. Δεν μιλώ καν για τα γενετικώ τροποποιημένα, ούτε τι ορμόνε. Οι Αμερικανοί τα χρησιμοποιούν για την ε, ανάπτυξη των ζώων. Τα αντιβιωτικά Ξέρουμε πόσο ε, κέριο είναι το θέμα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι το 70% των αντιβιωτικών που χρησιμοποιούνται στη ΣΥΠΑ χρησιμοποιούνται στα εκτροφία, στι κτηνοτροφικέ εκμεταλλεύσει, κατά τη ε, διάρκεια τη ανάπτυξη των ζώων με συγκεκριμένου στόχου. Ενώ το 10% χρησιμοποιείται μόλι για την θεραπευτική αγωγή και το 20% για, τα, ε, για του ασθενεί, του ανθρώπου. Μιλάμε για αριθμού που στην Ευρώπη δεν ε, στέκουν καθόλου. Εμείς κατά 70% ε, τη δική τους τη χρήση την απαγορεύουμε. Έχει απαγορευτεί από το 2006 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην ε, μιλήσω καν για το χλώριο που χρησιμοποιείται για την πλήση των σφαγίων πολιτικών, ούτε για το νερό. Στο, στην Ευρώπη χρησιμοποιείται μόνο πόσιμο νερό, στην Ιταλία ούτε καν αυτό. Διότι αμέσως μπαίνουν στο ψυγείο, και ε, ανεβαίνει η θερμοκρασία στο σημείο ακριβώ που πρέπει. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται δηλαδή είναι ακόμη πιο, ε, πιο αυστηρή. Για την ε, εξουσιοδότηση το είπαμε, για το γεωγραφικό εντοπισμό. Οι Αμερικανοί δεν αναγνωρίζουν τα σήματα. Εμείς έχουμε 271 στην Ιταλία. Τι άλλο να πω. Αυτό που ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εάν μπορεί αυτή την ε, μεθοδολογία να την αξιοποιήσει. Μια μεθοδολογία που την είχαμε υποδείξει εμείς. Να υπάρξει βέβαια αναγνώριση κοινέ προσεγγίσεις εκεί που υπάρχουν παρόμοια πρότυπα ή ιδάλλως να περιοριστεί η συνεργασία εκεί που συγκλίνουν εκεί μάλλον που είναι απομακρυσμένα μεταξύ τους τα πρότυπα να υπάρξει μόνο ανταλλαγή πληροφοριών ή εναρμόνιση προ τα ανώτερα πρότυπα. Διότι από αυτά που διαβάζω και καταλαβαίνω για το όλο θέμα, δεν νομίζω ότι αυτή την προσέγγιση έχετε προκρίνει. Για την επιστημιστική ασφάλεια, εάν δω το κεφάλαιο για τα φυτογειονομικά λόγου χάρη, εκεί δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ρύθμιση όπου να έχουν συναποφασίσει τα δύο μέρη της συμφωνίας, αλλά αμοιβαία αναγνώριση των αντιστοιχειών που θα μας επιτρέψει να αποδεχτούμε την νομοθεσία και των δύο πλευρών χωρίς να προστεθεί μια σφαιρική εξέταση, μια αναθεώρηση των κανόνων. Βλέπετε λοιπόν τι μπορεί να προκύψει σε, επίπεδο αποκλήσεων απόψεων, διαφωνιών. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει κάτι πιο συγκεκριμένο για αυτά τα θέματα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε η κυρία Ντορνανό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά το 12ο γύρο των διαπραγματεύσεων, που επικεντρωνόταν κυρίως στην ε, κανονιστική συνεργασία, φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα σύγκληση σε μερικά σημεία. Μπορείτε να μας πείτε πού εντοπίστηκε τέτοια σύγκληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαιώνει ότι ε, θα αποκλείσει από τις διαπραγματεύσεις αυξητικές ορμόνες και τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Πάλι καλά. Βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα ιχνηλασιμότητε. Γιατί στι Ηνωμένε Πολιτείε η ιχνηλασιμότητα εξασφαλίζεται για τα ε, ζώα που κυκλοφορούν μεταξύ των πολιτιών αλλά δεν ξεπερνάει το 18 μήνο έλεγχος, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει ε, διευρυμένο έλεγχο και μάλιστα από τη γέννηση. Και μάλιστα οι προδιαγραφές και τα πρότυπά μας ε, για την προστασία των ζώων και την καλή μεταχείριση επίση είναι διαφορετικέ. Υπάρχουν αντιφάσεις εδώ. Η ενημέρωση ήταν λυπή εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκρινίσει υπό ποιου όρου θα γίνουν όλα αυτά ή θα διευρύνει αυτούς τους όρους. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερο σημείο διαφορών. Αξιολόγηση κινδύνου για τι χημικέ ουσίε, για παράδειγμα η χημικά προϊόντα. Στις Πολιτείες μιλούμε για μη λογικό κίνδυνο, αλλά οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να εξετάζουν το κατά πόσο είναι ακίνδυνη μια ουσία. Επίσης, ε, παρόλο που υπάρχουν σοβαρές αφιβολίες για την μη επικινδυνότητα των προϊόντων, δεν απαγορεύεται αυτόματα η χρήση τους. Τι γίνεται λοιπόν με την αξιολόγηση κινδύνου. Υπάρχουν διαφορές εκεί. Τέλος, ε, στα θέματα της κανονιστικής συνεργασίας προβλέπονται κοινέ προδιαγραφές για τη διαχείριση του κινδύνου και αν ναι, ε, προς ποια μορφή και μεθοδολογία ανάλυσης οδεύουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σουίτσα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ παρακολουθώ επισταμένως εδώ και χρόνια αυτό το ζήτημα των διαπραγματεύσεων και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και οι συμπολίτε μου ενδιαφέρονται τα μάλα. Πολύ συχνά λαμβάνω μέρο σε εκπομπέ σε στρογγυλέ τράπεζε, όπου οι πολίτε θέτουν ερωτήσει. Αυτέ οι ερωτήσει σα μεταφέρω εδώ σήμερα και που ταλανίζουν του συμπολίτε μα. Εγώ δεν είμαι από τους πολέμιους του TTIP. Αντίθετα, είμαι υπέρμαχος του TTIP, είμαι υπέρ του TTIP. Θα ήθελα και στην ενία μας αγορά να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στις αγορές κυρίως της ΑΠΑ Ανατολής. Και γι' αυτό είμαι υπέρ του TTIP. Αλλά έχουν μείνει διευκρίνητες κάποιες ερωτήσεις. Η αξιοπιστία των διαπραγματεύσεων, η διαφάνειά τους, Φυσικά είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε τόσο σημαντικά και πλούσια ε, και πολυσέλιδα έγγραφα, αλλά ε, αυτή η αδιαφάνεια ενοχλεί τους Ευρωπαίους πολίτες που θα ήθελαν πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια για τόσο σημαντική συμφωνία. Μάλιστα Έχουμε χάρη στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάποιες βάσεις και κατευθυντήριες γραμμέ, αλλά εξακολουθούν να μένουν αδιευκρίνητες μερικές ερωτήσεις. Για παράδειγμα, προτείνεται νομοθετικές αλλαγές ε, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Χρειάζεται να αλλάξουμε και την κοινοτική νομοθεσία για να εγκριθεί αυτή η συμφωνία. Επίσης, πώς θα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υποβαστούν ή υποβαθμιστούν οι υψηλές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δύο είναι τα βασικά θέματα για τα οποία θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί κύρωση σε κάθε κράτος μέλος χωριστά και κύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν μας το είπατε ακόμη. Δεύτερο ερώτημα που βασανίζει τους πολίτες είναι αυτός ο μηχανισμός ISDS, Επίλυση διαφορών κράτους επενδυτή. Δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει συμφωνία για το θέμα αυτό. Αυτά τα δύο θέματα βασανίζουν κυρίως τους Ευρωπαίους πολίτες. Φυσικά ρωτάνε για την κλωνοποίηση, για τα φυτοφάρμακα, για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και ενδιαφέρονται να διαφυλαχθούν τηρηθούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές στα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ η κυρία Γκούτελαντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δώσατε για ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εγώ είμαι από τους συναδέλφους που ε, βλέπουν θετικά σημεία στο TTIP, αλλά χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις ε, και πολύ πιο μεγάλη ενημέρωση πριν λάβουμε τελική απόφαση. Πολιτική για τις χημικές ουσίες, αντιβιωτικά, ε, για τις γενετικώς τροποποιημένες οργανισμούς, φυτογειονομικά, δημόσια υγεία. Όπως είπε και η κυρία Μακίνας, θα πρέπει πριν να αποκρισταλώσουμε τη γνώμη μας, να είμαστε σίγουροι ότι το TTIP βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι θα είναι η οικονοποιητική έκβαση του ε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη γεωργία μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της χρήσης των φυτοφαρμάκων. Ήδη η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων ε, καταστρέφει τα οικοσυστήματα, τις μέλισσες, Αυτά όλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην πολιτική μας για τι χημικέ ουσίες. Εμεί προσπαθούμε να βελτιώσουμε και την προστασία του περιβάλλοντος και την δημόσια υγεία. Έχουμε την αίσθηση όμω ότι το TTIP άλλους σκοπούς επιδιώκει. Αν δεν καταφέρουμε να διαφυλάξουμε τις προδιαγραφέ και τα, πρότυπα, τα για την υγεία και το περιβάλλον, φοβάμαι ότι θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση στις διαπραγματεύσει. Θα πρέπει οι δεσμεύσει που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πολύ πιο σαφεί. Περιμένω τα αποτελέσματα και ευχαριστώ θερμά την Κομισιόν που ήρθε και μα παρουσίασε την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ, κυρία Εύη. Ε, ευχαριστώ. Και εγώ ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει κάποια πράγματα. Κατά πρώτον, ήθελα να κάνω μια διαπίστωση. Σήμερα μιλάμε ελάχιστα ακόμα, ιδιαίτερα στη χώρα μου την Ιταλία, σε επίπεδο κοινή γνώμη, ε, ευρέω κοινού, για το τι συμβαίνει με τι διαπραγματεύσει αυτέ. Γιατί είναι οι πρώτοι που θα υποστούν τι συνέπειε αυτή τη συμφωνία. Μια συμφωνία που βάζει στον μελετώνα τεκτύπου που έχουμε στη διάθεσή μα και έχουμε αναγνώσει τώρα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων βλέπουν ότι θα έχουμε αποτελέσματα σαφώ. Ε, πολύ απογοητευτικά σε σχέση με, τις, με τη βασική υποβάθμιση των προτύπων ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη υπόθηκαν πολλά από του συναδέλφου. Οι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν για πολυαριθμότατα από τα σημεία που όλο ιδιαίτερο άπτονται των αρμοδιοτήτων τη Επιτροπή αυτή. Εγώ όμω θέλω να κάνω μια ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ρήτρα του SDS. τη επίλυση διαφορών κράτο επενδυτού και του συστήματο που θα εφαρμοστεί. Είδαμε πρόσφατα την υπόθεση προσφυγή τη Καλιφόρνιας που θα ήθελε η γλυφοζάτη να ε, συμπεριληφθεί μεταξύ των ενδεχομένω καρκινογόνων ουσιών. Εδώ λοιπόν θα, ξέραμε, θα θέλαμε να ξέρουμε για μια τόσο, τόσο επικίνδυνη υπόθεση πώ θα μπορούσε να λειτουργήσει ο μηχανισμό απειλήση διαφορών ε, κράτου απέναντι απεντητή λόγου χάρη και τι θα συνέβαινε και στην περίπτωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση αν πρόκειται κάτι αντίστοιχο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα μετά από αυτή τη σειρά ερωτήσεων που έχουν ε, εκφραστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναδώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι απαντήσει του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που έθεσαν πολλά ερωτήματα. Να σας ομολογήσω ότι για έναν υπάλληλο αυτό μοιάζει με εξέταση. Ό,τι πιο κοντινό μπορώ να φανταστώ σε εξέταση. Να έρθω εδώ να σας προσπαθήσω να σας πείσω ε, να σας πείσω ότι παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τα σχόλια της Επιτροπής σας ε, εδώ και μήνες, από τότε που ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις αυτές μάλιστα. Να τονίσω λοιπόν αυτά που λένε οι βουλευτές, όλα αυτά έχουν ενταχθεί στις υπηρεσίες μας. Έχουμε 4-5 συναδέλφους εδώ πέρα από τα διάφορα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντιμετωπίζουμε τις ανησυχίες σας. Είναι καθήκον μας, είναι δουλειά μας να τα ενσωματώσουμε αυτά στον τρόπο εργασία μας. Να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει follow-up. Και θεωρώ ότι ο συνάδελφος Μπάλτσο, ο βουλευτής Μπάλτσο, μου ζήτησε μία ειλικρινή απάντηση στις ερωτήσεις του και πραγματικά με άγγιξε. Αλλά αυτό θα ήθελα να το κάνω σε όλους σας. Να ξεκινήσω με αυτά που με ρώτησε ο κ. Ντόρφμαν για το ερώτημα για, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις που υπάρχουν με τις εκλογές στη ΣΥΠΑ. Αυτό ασφαλώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαχειριστεί η αμερικανική πλευρά πιο πολύ του τουλεχθέντος, αληθεύει ε, βέβαια ότι οι δύο κορυφαίοι υποψέφοι στην Αμερική και ε, ο κύριος Τραμπ και η κυρία Κλίντον από πλευρά των Δημοκρατικών έχουν κάνει πολύ ξεκάθαρες δηλώσεις για την Αμερικανική εμπορική πολιτική, πιο πολύ σε ό,τι αφορά την ε, συμφωνία την διειρηνική, η οποία βρίσκεται ήδη σε φάση ε, υπογραφής αυτό ασφαλώς θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε, αλλά η κυβέρνηση είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το έργο το οποίο ξεκινήσαμε μαζί και όπως σας έχω πει και σε... στο παρελθόν θέλουν να ολοκληρωθεί εφέτος η διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το θέλει δυνατόν, αλλά τουλάχιστον αυτό έχουν δηλώσει δημόσια. Θυμάμαι μία συνάντηση πέρσι με τον κύριο Ντόρφμαν, ο οποίος μου εξήγησε ότι παράγει στην Αυστρία, στην περιφέρειά του, μήλα και εξάγεται ε, ο χυμός μήλου στην ε, Αμερική, αλλά όχι το ίδιο το μήλο, λόγω των ε, διαδικασιών που παίρνουν τόσο πολύ χρόνο. Θεωρούμε ότι αυτή η καταγγελία, αυτό αυτή η ένσταση είναι πολύ σωστή. Παίρνουν τόσο πολύ αγριοφρεκατικές διαδικασίες για τα τρόφιμα και τα λαχανικά και οι διαπραγματευτές μας συχνά υπενθυμίζουν στους Αμερικανούς πόσο παίρνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσαρμόσουν για να προσαρμόσουμε τις άδειες για τους γενετικά τροποποιημένους ε, οργανισμούς. Άρα οι Αμερικανοί παραπονούνται ότι μας παίρνει πάρα πολύ χρόνο να εγκρίνουμε γάματα μικρόν. Αλλά και εμείς απαντούμε ότι και αυτόν τους παίρνει πολύ χρόνο σε ό,τι αφορά και παράδειγμα τα μήλια, τα χλάδια, τη ρωσική αγορά. Ε, πριν από δύο χρόνια η Ρωσική Ομοσπονδία ξεκίνησε μια διαδικασία και ακόμα δεν έχουμε λάβει θετική απάντηση. Βλέπετε λοιπόν πόσο πολύπλοκες είναι αυτές οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης, γιατί έχουμε υπόψη όλες τις ανησυχίες που εκφράζονται από κάποιους από εσά ε, για το ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τις προδιαγραφές ασφαλείας μας. Αυτό το υποστηρίζει ακράδαντα ε, ο Επίτροπος, αλλά από την άλλη θα πρέπει να υπάρχει και μια δίκαιη πρόσβαση στις αλλαταπές αγορές. Και αυτός είναι ο στόχος των διαπραγματεύσεων πολύ το θέσατε αυτό το ερώτημα το, του, επίπεδου προστασίας. Δεν πρόκειται να πέσει το επίπεδο προστασίας μέσω του TTIP. Τα επίπεδα προστασίας, θα ήθελα να τονίσω, τα ορίζουν οι νομοθέτες, όχι οι διαπραγματευτές ε, της Γενικής Διεύθυνσης Trade. Εμείς ε, διευκολύνουμε τον μηχανισμό ρυθμιστικής συνεργασίας μεταξύ των νομοθετών και στις δύο πλευρές του εκλογικού, αλλά είμαστε απόλυτα κυρίαρχοι και το βλέπετε αυτό στο κείμενο του TTIP. Βλέπουμε ότι οι νομοθέτες θα εξακολουθήσουν να έχουν την επικυριαρχία τους σε ό,τι αφορά τα επίπεδα προστασίας. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν πρόκειται να δημιουργηθεί μια κοινή αγορά με τη ΣΥΠΑ όπως αυτή που υπάρχει με τα κράτη-μέλη, υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις ε, διαφορές. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε τη ρυθμιστική συνεργασία, προκειμένου να, μη, να μειωθούν τα απαραίτητα οι περαιτή στο εμπόριο. Να απαντήσω στον κύριο Στάς. Είναι, υπάρχει μία διαφορά Υπάρχει μια διαφορά λοιπόν μεταξύ των μη δασμολογικών φραγμών που αποτελούν μια ε, ε, διπλή αν θέλετε αλληλεπικάλυψη των φραγμών που είναι εις βάρος των εμπόρων μας και των παραγωγών μας και των φραγμών που είναι σημαντικοί για τους Ευρωπαίους ε, αλλά όχι απαραίτητα για τους Αμερικανούς. Και πολλοί από εσά το είπατε στα σχόλιά σας υπάρχουν σε, διάφορες, σε διάφορους τομείς διαφορετικές προσεγγίσεις και αυτό το διευκρινίσαμε και το διευκρινίζουμε στις διαπραγματεύσεις. Έχουμε πει ότι δεν διαπραγματευόμαστε τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την εισαγωγή βοήου κρέατος ε, που έχει υποστεί ορμονοθεραπεία, ότι δεν πρόκειται να το διαπραγματευτούμε. Είμαστε πάρα πολύ σαφείς ε, και υπάρχουν σαφέστατες παράμετροι που έχουν δημοσιευτεί σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσει Έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό δεσμευόμαστε. Φαίνεται αυτό και από το κείμενο που υποβάλαμε. Το κείμενο αυτό είναι στην διάθεσή σας. Όλες αυτές οι προτάσεις λοιπόν μπορούν να τις εξετάσουν οι βουλευτές στο σχετικό, στη σχετική αίθουσα ανάγνωσης και συμπεριλαμβάνεται και η αμερικανική πρόταση. Οι δικές μας προτάσεις δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Για όσους λένε λοιπόν ότι οι διαπραγματεύσεις είναι μυστικές και απόρριτες, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εδώ και πολλούς μήνες έχουμε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο τις προτάσεις μας και οι αιρετοί εκπρόσωποι μπορούν να πάνε και να βήμα παραπέρα, να έχουν πρόσβαση στον οποίημένο κείμενο που περιλαμβάνει και τις αμερικανικές προτάσεις και αυτά διατίθενται από τα Χριστούγεννα και μετά και στα εθνικά κράτη-μέλη. Υπάρχουν 23 κράτη-μέλη τα οποία ως τώρα, 23 λοιπόν, έχουν δημιουργήσει τέτοιες αίθουσε ανάγνωσης εθνικές για να μπορούν να συμβουλευτούν και οι εθνικοί βουλευτές τα ενοποιημένα κείμενα. Όχι μόνο εσείς λοιπόν ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και οι συνάδελφοί σας από τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν πρόσβαση στα ενωπημένα αυτά κείμενα και μπορείτε φυσικά να μας θεωρείτε και να μας καλέσετε ως υπεύθυνου σε περίπτωση που υπάρχουν κάποια τμήματα ε, στο κείμενο αυτό τα οποία θα φέρετε να τα θέσετε ένα φιβολό Επίσης, να αναλύσω κάποια από τα σχόλια που πολλοί από σας έκαναν και να απαντήσω όσο πιο δικαιωτικά γίνεται. Για την ερώτηση του κυρίου Μπαλάς για την ε, μελέτη δικτύπου και την ε, μελέτη ε, εφικτού εδώ η έκθεση θα γίνει από επιχείρηση ανεξάρτητη, τελείως αυτόνομα η επιχείρηση λαμβάνει γλώσσα όλων των κεφαλαίων που θα πρέπει να μελετηθούν και θα έχει και ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Στόχος της έκθεσης που θα ξεπερνάει τις 100 είναι να κάνει μια ποιοτική αποτίμηση αλλά και ποσοτική για τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας τη στιγμή που θα αρχίσει να υλοποιείται. Η μελέτη στρέφεται και μελετά και συγκεκριμένους τομείς όπως για παράδειγμα τα κοινωνικά δικαιώματα ή ο τομέας των ναυτιλιακών, της ναυτιλίας, έχουν εντοπίσει δέκα τουλάχιστον τομείς όπου όλα αυτά βρίσκονται κατά την άποψή τους στην καρδιά μιας ε, ε, sustainability impact assessment όπως λέγεται, δηλαδή μελέτη αντικτύπου βιωσιμότητας και μεγάλη ε, έμφαση στην ποιοτική διάσταση αυτής της έκθεσης. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να έχουμε μια συμφωνία στο δυνατόν καλύτερη από ποιοτική άποψη. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι απλώς να απελευθερώσουμε την αγορά, αλλά η συμφωνία αυτή είναι μια εντολή τροποντινά για να προάγουμε κάποιες δικές μας αξίες, ακόμη για να υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Όμως, οι διαφορές ΗΠΑ Ευρώπης είναι πιο μικρές εάν συγκρίνουμε λόγω χάρη τι συμβάνει με άλλους εμπορικούς μας εταίρους, όπως η Ινδία, η Βραζιλία, η Κίνα ή η Ομοσπονδία της Ρωσίας. Επίσης για τις ερωτήσεις της κυρίας Μίλλερ για τις ομάδες πίεσης, το lobbying. Να πω ότι έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις ε, στο κείμενο για την βιωσμένη ανάπτυξη που είχαμε υποβάλει και σε εσά το Δεκέμβριο. Και εκεί περιλαμβάνονται δεσμεύσεις για τη βιώσιμη συντήρηση της δασοκομείας, για την υλοτομία, την παράνομη υλοτομία και την χρήση ε, συγκεκριμένων κανόνων για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών από, το μηχανικό μας ε, κλάδο, καθώς και ε, το τι θα γίνει με τις ανάλογες σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Αυτά είναι γνωστά και στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων TTIP. Για τον κύριο Στάς, και τις ερωτήσεις του. Νομίζω ότι εν μέρη ήδη έκανα την διάκριση για τις μη δασμολογικούς φραγμούς που πολλές φορές έχουν να κάνουν με το πώς εκφραζόμαστε απέναντι σε διαφορές του πολιτικές στάσεις. Θα παραμείνουν διαφορές και μετά την επίτευξη συμφωνίας ενδεχομένως. Η συμφωνία τύπου σκοπό δεν έχει να δηλήσει αξίες που προωθούνται ή στηρίζονται από το Συμβούλιο και που έχουν ε, εκφραστεί και παγιωθεί σε κείμενα των θεσμικών οργάνων μέσα από μια σειρά ετών. Όμως, ό,τι φορά την εφαρμογή της συνθήκης, την αμοιβαία αναγνώριση, την αντιστοιχία λόγω χάρη, αυτό και πάλι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να το δει και να το εξετάσει δεν είναι κάτι που θα το χάσετε ή θα σας το κρύψουμε στα πλαίσια μιας αδιαφανούς γραφειοκρατικής διαδικασίας. Για το πρόγραμμα REACH νομίζω ότι σωστό είναι να πούμε ότι προς τη υπάρχει διαφορά στην προσέγγιση μας μεταξύ μόνο και των ε, Αμερικανών φίλων μας, αλλά έγινε και ένα σχόλιο για τις επενδύσεις. Ο κύριος Τάστο ρώτησε το θέμα αυτό, ο κύριος ε, το που έχουμε φτάσει με αυτό το τόσο σημαντικό μέρος των διαπραγματεύσεων. Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα εδώ στο Κοινοβούλιο αυτά έχουν συζητηθεί επί μακρόν, αλλά και σε επίπεδο κοινή γνώμη, με αντικρουόμενε απόψει και διαφωνίε για το τι γίνεται στι διαπραγματεύσει TTIP. Μετά από μακροσκελέστατε διαπραγματεύσει με συμμετοχή των ενδιαφερομένων τη κοινωνία των πολιτών, με μακροσκελεί συζητήσει εδώ, με συζητήσει με τα κράτη-μέλη, που να θυμίσω είναι η βασική ε, υπεύθυνη για τέτοιου είδου ε, συμφωνίε, έχουμε νέα πλατφόρμα για την ε, επίλυση διαφορών δεν είναι καμιά επαναστατική αλλαγή σε σχέση με το παλιό ISDS, το Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών Κράτους Επενδυτή. Απλώς τώρα προτείναμε να ε, στηριχθεί η δικαστική διάσταση της ε, επίλυσης επενδυτικών διαφορών. Και αυτό για να υπάρξει και συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτό επισήμως αναγνωρίζεται στο κεφάλαιο της, ε, του μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτικού κράτους. Η δικαστική λοιπόν διάσταση σημαίνει ότι τα μέρη που ε, είναι μπροστά στο δικαστήριο ως ότι οι διαιτητές στα δικαστήρια θα κριθούν από δικαστές εθνικούς οι οποίοι ανεξαρτήτως και τυχαία θα διοριστούν για να εξετάσουν αυτή την υπόθεση με πλήρη διαφάνεια, δημόσιας ακροάσεις και δυνατότητα έφεσης. Αυτό σε συνδυασμό με ρητή ε, τεκμηρίωση του δικαιώματος του ρυθμίζει είναι κατά την άποψή μας η κατάλληλη απόκριση για να ξέρουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των ε, εργαλείων και των πολύ έντονων απόψεων που εξέφρασε η κοινωνία των πολιτών σε σχέση με το θέμα. Βεβαίω, αυτέ είναι διαπραγματεύσει. Για την ώρα αυτή είναι η δική μα πρόταση. Περάσαμε τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων στι συζητήσει μα με του Αμερικανού μα εταίρου να εξηγούμε γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η σωστή ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί και ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί για του Ευρωπαίου. Δεν είναι μυστικό. Το είπαμε και είναι και μια άποψη ακλόνητη του δικού σας του σώματος για την προστασία των ε, επενδύσεων του τελευταίου μήνες, τα είπατε, και ξέρουμε ότι όλα αυτά στο τέλος έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να τα εξετάσετε εσείς για να τα εγκρίνετε. Ο κύριος Πότς άρεσε, ρώτησε κάποιες ερωτήσεις για, την, ε, για το απόρριτο. Για την πρόσβαση λοιπόν στα κείμενα, ρωτήσατε επιπλέον τι γίνεται με την ενδεχομένω ασυμμετρική φύση, τον ασυμμετρικό χαρακτήρα αυτή τη συμφωνία. Είναι σαφέ ότι οι ΗΠΑ είναι χώρα ομοσπονδιακή. Όμω σε πολλέ περιπτώσει και σε πολλού τομεί πολιτική στην Ευρώπη είμαστε και εμεί ομοσπονδοποιημένοι. Μπορούμε λοιπόν και ισότιμα να αντιμετωπιστούμε με του Αμερικανού. Δύο οικονομίε που έχουν περίπου το ίδιο μέγεθο και το ίδιο επίπεδο ανάπτυξη μπορούν να συνεργαστούν, απλώς αυτό εξαρτάται από τη δυνατότητα να είμαστε ενιαίος κάτω μέλος. Το Αμερικανικό Κοινοβούλιο είναι το άλλο θεσμικό όργανο που θα αποφανθεί επί τη συμφωνία. Θα πρέπει λοιπόν να αποστέλουμε διαρκώ μηνύματα για την ανάγκη εξέβρεση ισορροπία στην τελική συμφωνία. Αυτό είναι κάτι που από την πλευρά του Συμβουλίου βρίσκεται στο επίκεντρο των μεριμνών τους ε, και πολλά κράτη-μέλη στρέφουν το βλέμμα σε αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο των δημοτεύσεων. Χρειάζεται ισορροπία, υψηλά πρότυπα και διεξοδικότητα στο να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα για τους πολίτες μας ώστε να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής από την ευρωπαϊκή πλευρά σημαίνει ότι θα γίνει πολλές φορές με κατεξουσιοδότηση πράξης και βεβαίως το σώμα σας ότι κι θα τις δει. Σε ό,τι αφορά το υπο επίπεδο, το πολιτιακό επίπεδο στι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πολύ θέσατε σχετικό ερώτημα. Από τη στιγμή που συναυθεί η TTIP συμφωνία και κυρωθεί και από τις δύο πλευρές, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναλάβει την ευθύνη για την εφαρμογή της συμφωνίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Και πρόκειται για μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει δεσμευτικούς μηχανισμούς για την επίλυση διαφορών σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι δεσμεύσει σε πολιτιακό επίπεδο. Οπότε μπορούμε να πάμε και στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν υπάρχουν τομεί πολιτική που εμπίπτουν στι αρμοδιότητε των πολιτιών στι Ηνωμένε Πολιτείε Όπως και εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλού τομεί που δεν εμπίπτουν στι κοινοτικέ αρμοδιότητε, αλλά είναι εθνικέ αρμοδιότητε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το πολιτιακό επίπεδο, το θέμα είναι τι δεσμεύσει εμεί μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ σε τομεί που η αρμοδιότητα ανήκει σε πολιτιακό επίπεδο, στις πολιτείες, σε πολιτιακό επίπεδο, υπομοσπονδιακό δηλαδή. Επίσης, τα θέματα των δημοσίων συμβάσεων. Εκεί έχουμε πολλές ε, ε, διακρίσεις εις βάρος ε, των Ευρωπαίων. Και τα περισσότερα θέματα αυτά εγκρίνονται και εφαρμόζονται σε πολιτιακό επίπεδο. Οπότε θα πρέπει στις ε, διαπραγματεύσεις για τις κρατικές προμηθείς της δημόσιες συμβάσεις να βρούμε δεσμεύσεις που θα μπορέσουν να τις αποδεχθούν και οι πολιτείες ε, και οι πόλεις ε, και σε υπόμοσποδιακό επίπεδο. Το ίδιο ισχύει και για την αναγνώριση των προσόντων. Και αυτό είναι αρμοδιότητα των πολιτιών. Και εμείς έχουμε μια αγορά, αλλά παρόλα αυτά σε πολλούς τομείς ε, έχουμε αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οπότε με το διαπραγματεύσεων ε, είναι και η ανέβρεση σωστής ισορροπίας και ισορροπίας μεταξύ των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται σε ε, ομοσπονδιακό επίπεδο και εκεί που υπάρχουν αρμοδιότητες των πολιτιών να, δούμε, να εξασφαλίσουμε δέσμευση και των πολιτιών ώστε να έχουμε κάποια αποτελέσματα που θα είναι δεσμευτικά στη συνθήκη, στην συμφωνία αυτή την TTIP. Και από τη στιγμή που γίνουν αποδεκτές αυτές οι δεσμεύσεις και αποκρισταλωθούν σε δίκαιο, στη συμφωνία, θα πρέπει να γίνουν σεβαστές και σε επίπεδο πολιτιών. Το αμερικανικό σύστημα είναι πολύ διεξοδικό σε ό,τι αφορά, όπως ξέρετε, την ε, εφαρμογή. Ο, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις κυρίας Γκέρλινγκ, προσπαθούμε και καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες ε, να εκπονήσουμε τέτοια κείμενα και να ενοποιήσουμε μερικά από αυτά. Οπότε μέχρι το καλοκαίρι εσείς και τα κράτη-μέλη θα είστε σε θέση να ε, διαπιστώσετε τι προσέγγιση υιοθετήσαμε στους επιμέρους τομείς. Και φυσικά υπάρχουν διαφορές. Αλλιώς αντιμετωπίζουμε εμείς ε, τα χημικέ τις χημικές ουσίες και αλλιώς τα, ε, τα φάρμακα που απαιτούνται επιθεωρήσεις ε, των εργαστηρίων ή αλλιώς αντιμετωπίζουμε τα οχήματα, την κατασκευή οχημάτων. Και επίσης υπάρχουν διαφορές που είναι το αποτέλεσμα εύλογων πολιτικών επιλογών. Μεταξύ αυτών και των επιλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί που υπάρχουν τέτοιες διαφορές και χάσματα, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή, θα τα αποδεχθούμε. Εκεί όμως που υπάρχουν διαφορές που δεν έχουν νόημα σε τη φορά την ε, παροχή ασφάλειας για τους πολίτες. Για παράδειγμα, να μην υποβαθμίζεται η ασφάλεια ε, όταν ε, χρησιμοποιούμε ένα αμερικανικό αυτοκίνητο ή ένα ευρωπαϊκό. Αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Βέβαια, κυρίως ε, ευρωπαϊκές είναι αυτοκινητοβιομηχανίες. Ε, βέβαια, αυξάνεται το κόστος όταν υπάρχει επικάλυψη και μάλιστα περιττή επικάλυψη νομοθετική. Και τμήμα της κανονιστικής συνεργασία είναι να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των νομοθετικών αρχών, ώστε το επίπεδο προστασίας να αναβαθμιστεί και σε καμία περίπτωση να μην υποβιβαστεί. Επίσης, ε, εκεί που έχουμε παρόμοια θέματα, όταν ε, κάνουμε μια αναβάθμιση, επειδή έχουμε καλύτερη πρόσβαση στην επιστημονική έρευνα, γιατί είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε κανονιστικό επίπεδο ε, ή αν μπορούμε να διαθέτουμε στην αγορά γενώσιμα φάρμακα πολύ πιο γρήγορα, ώστε να έχουμε προσιτά φάρμακα σε προσιτές τιμές για τους πολίτες, χάρη στην ε, επιτάχυση της διαδικασίας έγκρισης, νομίζω ότι αυτό είναι προς όφελος των συμπολιτών μας. Κυρία Γιατανμάκη, μιλήσατε και ρωτήσατε για, τις, για τους δασμούς. Προχωρούμε και έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Ε, βρισκόμαστε σχεδόν στην τελική φάση ε, της συμφωνίας για τους δασμούς. Τώρα, που έχουμε προβλήματα. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Υπάρχουν όντως μερικοί τομείς ε, στις διαπραγματεύσεις που είναι πιο δύσκολοι και ο δρόμος μακρύς ακόμη. Και αφορούν κυρίως ε, την πρόσβαση στις αγορές, που είναι το ψωμοτήρι των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Και το βλέπετε και από τις μέχρι τώρα εμπειρίες η σωστή ισορροπία, η σωστή προσέγγιση στα θέματα των υπηρεσιών, των δημοσίων συμβάσεων, εκεί είναι που είναι δύσκολη, σκληρό καρύδι το θέμα της πρόσβεσης της αγορές και το θέμα του ανοίγματο των αγορών και για τους μεν και για τους δε. Η κυρία Ντονάνο μίλησε για την ιχνηλασιμότητα. Όντως υπάρχουν ε, διαφορές και σε αυτό το θέμα και στην καλή μεταχείριση των ζώων. Αλλά σε πολλούς από αυτούς τους τομείς προσπαθούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Μπορεί να μην είναι επαναστατική, να μην είναι σούπερ εντυπωσιακή, αλλά δείτε την πρόοδο που έγινε για την καλή μεταχείριση των ζώων, για τη χρήση των αντιβιωτικών, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς που αφορούν τις αρμοδιότητες και τα ενδιαφέροντα της δικής της Επιτροπής διαπιστώνεται ότι προσπαθούμε να σημειώσουμε πρόοδο με τους ε, Αμερικανούς αντισυμβαλλομένους. Και σε ό,τι αφορά την ε, εκτίμηση κινδύνου, αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της κανονιστικής συνεργασίας και η υπέρτερη αρχή είναι ότι αποφασίζουν οι νομοθέτες και όχι οι διαπραγματευτές. Οι νομοθέτες αποφασίζουν σε τι βαθμό θα προβλέψουν μηχανισμούς ε, ή υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί για την αναγνώριση της ισοδυναμίας. Και τέτοιοι μηχανισμοί θα υποβληθούν προς εξέταση ως ονοπο, είτε στα πλαίσια της συμφωνίας είτε μετά. Πάντως θα είμαστε πολύ διεξοδικοί εδώ. Σε ό,τι αφορά τη γλυφοσάτη και τα φυτοφάρμακα, νομίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την έγκριση στο σημείο αυτό και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Ελπίζω να εξάντλησα τις ερωτήσεις. Ε, δεν ξέρω αν πέρασα τις εξετάσεις ή έμεινα μεταξυταστέως. Πάντως προσπάθησα να σας απαντήσω. Και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε τις προτάσεις σας είτε δημερός είτε με επιστολές στα γραφεία μας ε, και πρόθυμοι να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσεις της. Είμαι πεπισμένος ότι η Επιτροπή αυτή θα παρακολουθήσει προσεκτικά όλη την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων TTIP και τώρα περνάμε στο σημείο 6. Προετοιμασία τη μετακυκλογική αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η συμβολή του Κοινοβουλίου ανάψη τη πρόταση τη Επιτροπή. Παρακαλώ όσοι θέλετε να φύγετε, εάν μπορείτε ησύχω, Εάν θέλετε Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνετε πηγαδάκια, κάντε το έξω, εκτός σας παρακαλώ. Και ευθύ αμέσω να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, στον Φράνσις Γκάμπους από το ΕΛΚ. Θα μπορούσατε φίλοι μου να φύγετε ησύχως από την αίθουσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του στην Ολομέλεια του Στρασβούργου παρουσιάζοντας ε, τις κατευθυντήριες γραμμές για ε, τη δράση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη θητεία ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προσανατολίσει τον ε, κοινοτικό προσανατολισμό προς θέσεις απασχόλησης, οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Έτσι και με αυτά τα κριτήρια εκπώνησα και εγώ το σχέδιο Έκθεση, που είναι το αντικείμενο τη σημερινή συζήτηση και για το οποίο περιμένω τη συνεργασία με τι πολιτικέ ομάδε και του και ηγητές για να το βελτιώσουμε. Προσπάθησα πάντως να κρατήσω ισορροπίε ε, στο πρώτο σχέδιο αυτού του εγγράφου. Πολλές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για το περιβάλλον και θα πρέπει να προσαρμόσουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στρατηγική για το 2020. Συγγνώμη, μια στιγμή κύριε Σιγητά. Παρακαλώ τα πηγαδάκια είπαμε εκτός εθούσης. Συνεχίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πολλές οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Πάντως ε, θα πρέπει να προσαρμόσουμε και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στη στρατηγική για το 2020 για να υλοποιήσουμε τους στόχους ε, ε, του Παρισιού στην διάσκεψη COP21. Οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν ουσιαστική απειλή για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να τι μετριάσουμε ώστε να αφήσουμε σωστή παρακαταθήκη σε επόμενες γενιές. Επίσης να διαφυλάξουμε τη βιοποικιλότητα και να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη. Ο πλούτος μας έχει πολλές πηγές, ιστορία, κουλτούρα, πολιτισμό, θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων με την οικονομική ανάπτυξη. Δεν είναι αντιφατικές αξίες μεταξύ τους. Επίσης, ε, κυκλική οικονομία. Ε, γιατί για να εξασφαλίσουμε την επιβίωση του πλανήτη μας θα πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα συμβατά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης ε, για να εξασφαλίσουμε μια ευημερία που θα πρέπει να είναι προσιτή σε όλους τους πολίτες. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία. Αυτή είναι η πρόκληση. Το πρόγραμμα LIFE, όπως λέει και το σχέδιο έκθεσης, αντικατοπτρίζει ε, αυτά τα τρία, αυτές τις τρεις αξίες που μας είπε και ο κύριος Γιουνκέρ. Ε, εργασία με προσθέμενη αξία, οικονομική ανάπτυξη, καλύτερο μέλλον. Το LIFE είναι ένα παράδειγμα, αλλά έχουμε και άλλα αναπόφευκτα προγράμματα, πολύ σημαντικά, με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τα χωροκατακτητικά είδη που έχουν επιβλαβεί επίδραση στο σύστημα και χρειαζόμαστε διάστατες προσεγγίσεις για να τα καταπολεμήσουμε ε, με συνδυασμό διαφόρων πολιτικών, περιβαλλοντική υγεία και ούτως άλλως και, και ούτω καθεξής. Τα χωροκατακτητικά είδη σημαντική απειλή θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε με πυγμή και το θέμα αυτό και να διαθέσουμε πόρους για να διαφυλάξουμε την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Επίσης, ε, το πρόγραμμα για την ανάπτυξη, ε, Health for Growth, υγεία για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δημογραφικές προκλήσεις και όπως είδαμε στα τέλη του 2014 και στις αρχές του 2015 δεν ζούμε σε, μια, σε ένα απομονωμένο νησί μακριά από τα προβλήματα του κόσμου. Είχαμε την επιδημία του έμπολα, σήμερα έχουμε τον ιό Ζήκα, δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους για να αναχαιτήσουμε αυτές τις απειλές και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ποιοτικά συστήματα υγείας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Εν κατακλείδη, να αναφερθώ σε, στο τελευταίο σημείο που περιλαμβάνει ε, η γνωμοδότησή μου, πολύ σημαντικό όμως. Τα χρόνια της κρίσης, ε, όπως μας λένε οι μελέτες, άφησαν όχι μόνο μεγάλες οικονομικές ανισότητες, αλλά και ε, κλάδεψαν την αγοραστική δύναμη πολλών ευρωπαϊκών οικοκυριών. Έχουμε ακόμη και πρόβλημα υποσυτισμού ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους και τους ηλικιωμένους εξαιτία ε, των περίκοπων των συντάξεων. Θα πρέπει λοιπόν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να προβλέψει τους απαραίτητους σπόρους για να καταπολεμήσουμε τον υποσυτισμό σε όλες τις ηλικίε. Επίσης, ε, θα πρέπει με την ενδιάμεση αναθεώρηση όχι μόνο να, να προσανατολίσουμε τον προϋπολογισμό μας ε, για περισσότερες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, αλλά και για την ενίσχυση της ευημερίας μας. Αυτό είναι, επαναλαμβάνω, το πρωτόλιο σχέδιο. Περιμένω τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών και των, των μελών των πολιτικών ομάδων για να το βελτιώσω και να το εμπλουτίσω. Ευχαριστώ κύριος Γραμματικάκης από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι χαρά μου γιατί η εισήγηση του κυρίου Καμπής έχει εύστοχα εντοπίσει τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα πρέπει να ανταποκριθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Θα ήθελα απλώ και εγώ με τη σειρά μου να τονίσω κάποια σημεία για τον προβληματισμό το γενικό σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα δεδομένα όπως ξέρουμε όλοι στην περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία έχουν αλλάξει. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή και βέβαια το δικό μας ευρωπαϊκό πακέτο για τη μείωση των ρήπων όπως και την ομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρήπανση και βέβαια ακόμα πιο σημαντικό για την κυκλική οικονομία. Λόγω και της οικονομικής κρίσης, όπως ανέφερε και ο εισηγητής, δυστυχώς η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας είναι, φοβόμαι να το πω, αποσπασματική και ελλειπής. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι βέβαια το πρόγραμμα LIFE Δεδομένου λοιπόν των νέων αυτών συνθηκών είναι πιστεύω σκόπιμο να διερευνήσουμε τρόπους τους πιο θα έλεγα αποδοτικούς για να στηρίξουμε το πρόγραμμα αυτό όσο τουλάχιστον μπορούμε. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα της χρηματοδότησης για το κλίμα σε δύο επίπεδα. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο όπου θα έχουμε νέους στόχους για το 2030 και σε παγκόσμιο βέβαια επίπεδο με τη Συμφωνία του Παρισιού η οποία προβλέπει όπως γνωρίζετε χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών σε ύψους 100 δις δολαρίων ετησίως. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο η στροφή προς μια βιώσιμη οικονομία, ελεύθερη βέβαια από εκπομπές άνθρακα, είναι πάγιο έτοιμο. Ίσως λοιπόν η αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι μια ευκαιρία για να διεκδικήσουμε την αύξηση του ποσοστού 20% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που έχει συμφωνηθεί ότι θα χρηματοδοτεί έργα και πολιτικές σχετικά με το κλίμα. Στο παγκόσμιο επίπεδο τώρα θα πρέπει προς το παρόν να κρατήσουμε μια στάση αναμονής, έτσι πιστεύω, έως ότου αποσαφινιστεί πώς θα καταμεριστεί το ποσό των 100 δις ο προϋπολογισμός θα πρέπει να παίξει το ρόλο που του αναλογεί, κυρίως από τους πόρους για την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά θα πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί, ώστε τα κράτη-μέλη να μην ρίξουν τις δικές τους ευθύνες στον προϋπολογισμό εις βάρον άλλων προγραμμάτων και πολιτικών. Και εδώ χαίρομαι ε, να αναφερθώ σε αυτό που τόνισε ο κύριος συζητητής, ότι η οικονομική κρίση έχει φέρει προβλήματα ακόμα και επισητισμού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στη χώρα μου την Ελλάδα. Τέλος, ένα σχόλιο για το ζήτημα των ιδίων πόρων. Εγώ το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αγνοήσουμε ως Επιτροπή τη συζήτηση σχετικά με την εξέβρεση ιδίων πόρων. Πρέπει να εξετάσουμε και να προτείνουμε λύσεις στη βάση της αρχής ο Ριπένον πληρώνει. Πολύ απλό αλλά πολύ σημαντικό. Έτσι διεκδικούμε όχι μόνο γνήσιους ιδίους πόρους αλλά και συνέργειες με την περιβαλλοντική και κλιματική μας πολιτική. Σε αυτά τα μεγάλα θέματα περιμένω κύριοι συνάλφοι και κύριοι συγητά τη συνεργασία όλων σας. Ευχαριστώ πολύ. Η Julie Gerling από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Ναι, κάποιες γενικές παρατηρήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην ομάδα μου πιστεύουμε ότι κανένα λογικό οργανισμό δεν προβλέπει προπολογισμό για 5-6 χρόνια χωρί να κατανοεί ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και προσαρμογή αυτού του αρχικού προγραμματισμού. Όμω, επιμένουμε ότι για τα συνολικά ποσά που θα εκταμιευθούν δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ε, νέα δεδομένα για αύξηση πόρων. Δεν συμφωνώ καθόλου αυτό. Το θέμα είναι τι θα πρέπει να κάνουμε με όσα έχουν διαθέσει τα κράτη-μέλη σε συμφωνία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Αυτό που λέμε εμείς λοιπόν είναι ότι τα συνολικά επίπεδα δαπανών δεν πρέπει να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση, αλλά αυτό που πραγματικά παροτρύνουμε να γίνει είναι να υπάρξει μια ψύχρεμη και προσεκτική εξέταση για το τι γίνεται στα διάφορα χαρτοφυλάκια του πολιετούς δημοσιονομικού. Διότι ακριβώς τον προπολογισμό μας, περισσότερο από κάθε άλλον οργανισμό στον οποίο εργάστηκα ή από την εθνική μας κυβέρνηση, Έχουμε μια σειρά από ιερές αγελάδες που φαίνεται ότι δεν μπορούμε να τις ακουμπήσουμε καθόλου. Ασχέτως των, ε, της των γεγονότων, όπως η αυξανόμενη σημασία των κλιματικών αλλαγών ή των θεμάτων των προσφύγων. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν για το πώς ε, προγραμματίζονται τα κονδύλια του προπολογισμού. Πρέπει να δούμε κάποιους από τους τομείς που θεωρούμε ότι είναι άθικτοι, ανέγκυχτοι. Δεν πρέπει να ισχύει αυτό. Δεν σημαίνει ότι αμφισβητώ το 20% του προπολογισμού που έχει συμφωνηθεί στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαίσιου για τη δράση αναχέτηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό το βρίσκω απολύτω εύστοχο. Αλλά πρέπει να δούμε πού ακριβώ κατευθύνονται τα κονδύλια και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα δαπανούμε συνετά, ώστε να, ε, ακριβώς να πετυχαίνουμε τους στόχους που αρχικά έχουμε ορίσει. Ε, συνοπτικά, πιστεύω ότι σε αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε τα σωστά ποσά ήδη και πραγματικά θα ήθελα να γίνει μια τολμηρή συζήτηση για τις δεσμεύσεις μας, για το πώς δαπανούνται τα ποσά αυτά, αλλά χωρίς καμία απόπειρα για το συνολικό χαρτοφυλάκιο του 2013 να υπάρξει αλλαγή. Ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί εκείνη η συμφωνία και θα ήθελα να παραμείνουμε πιστοί σε αυτήν. ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ο κύριος Τορβάλτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. με τους διάφορους δημοσιονομικούς περιορισμούς βρισκόμαστε στο κέντρο των προβληματισμών μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές τις μέρες. Ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς όσο και να έχουμε επικοδομητική προσέγγιση. Συνήθως τα προβλήματα τα εξετάζουμε με τις καλύτερες των προθέσεων. Όλοι μας ταυτόχρονα γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο μπορούν να μας πάνε μακριά οι καλές προθέσεις κάποιες φορές. Η καλή πρόθεση συνήθως δεν αρκεί. Χρειάζονται και δράσεις, πράξεις, για να μεταφραστούν και αυτού του είδους οι προσανατολισμοί σε συγκεκριμένα γεγονότα. Ο στόχος μας με το χαρτοφυλάκιο αυτό ή με τη συζήτηση αυτή καλύτερα είναι να βοηθήσουμε την Επιτροπή Προπολογισμών να ε, Πιλοτάρει όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Γι' αυτό θα προτείνω ορισμένε συγκεκριμένε τροπολογίε και θα ήθελα να κάνω έκκληση για να θεώρηση του πολιτή νομοσυνομικού πλαισίου εν ώψη τη συμφωνία των Παρισιών και το άρθρο 19 του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου το διευκρινίζει αυτό. Χρειαζόμαστε και νέου κανόνε για τα διαφορετικά ταμεία ώστε να διευκολύνουμε τη λειτουργία του και να εξυπηρετήσουμε του κλιματικού μα στόχου Πρέπει επίση να ξαναδούμε το επίπεδο των ε, δεσμεύσεων με έναν αποτελεσματικότερο μηχανισμό εξετασής και αναθεώρησης. Επίσης, σημαντικό είναι να γνωρίζουμε γιατί υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ιδίως στα περιβαλλοντικά προγράμματα. Οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν προβλήματα στον τομέα των περιβαλλοντικών μας προτεραιοτήτων. Επίσης θα θυμάστε τι δυσχερείς συζητήσει είχαμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων. Πρέπει να δούμε πώς οι περικοπές στο Horizon 2020, το ορίζοντα 2020, επηρεάζουν τα πράγματα. Υπήρξε μια μετατόπιση κονδυλίων από το Horizon 2020 προς το ΕΦΣΥ, αλλά ο αντίκτυπος στο περιβάλλον μπορεί να είναι σημαντικός. Αυτές είναι οι βασικές μου ερωτήσεις και Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την αναμενόμενη καλή συνεργασία που θα έχουμε και για τις αλλαγές που επιφέρει. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, no. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιο θέλει το λόγο. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Όχι, κυρία Πύρη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, όταν ε, συνήψαμε τη συμφωνία για το κλίμα, στην Ολλανδία ήμασταν πάρα πολύ θετικοί και ήταν θετικοί και ε, οι επιχειρηματίες. Ε, πιστέψαμε ότι θα ήταν θετικό, ότι θα φέρει πολλές θέσεις εργασίας, αλλά να δούμε τι έχει γίνει τελικά. Η ερώτηση που έγινε, κοιτάμε και το ΕΦΣΗ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά το πριν δεν είναι σαφές Πού θα πρέπει να πάει κανεί, πού θα πρέπει να απευθυνθεί. Αυτό δεν ξέρουν πολλέ επιχειρήσει και θα πρέπει να το ευκρινίσουμε. Κάτι άλλο. Κατέθεσα μια σχετική τροπολογία. Όλοι οι τομεί θα πρέπει να έχουν ίση αντιμετώπιση και μεταχείριση. Ευχαριστώ τον εισήγητη για την ε, προσέγγιση του. Έχουμε ανταγωνιστικέ θέσει μεταξύ χωρών. Ένα παράδειγμα. Στην Ολλανδία, κατά το ίμιση, οι αγροτικέ επιχειρήσει έχουν σχεδόν πτωχεύσει, γιατί έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην ευημερία των ζώων, σε περιβαλλοντικά πρότυπα, αλλά σε ό,τι αφορά την τιμή στην αγορά δεν ε, τα βγάζουν πέρα τελικά. Και θα ήθελα να αναφέρω και το Natura 2000. Πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά. Πρόσφατα εδώ στο Κοινοβούλιο αποφασίσαμε τι θα κάνουμε και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αλλά οι αγρότες λένε τελικά τι θα γίνει με τα δικά μας ε, τα πράγματα και μιλάμε για ε, οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ήπεθρο. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε περιθώριο σε αυτούς ανθρώπους για να πετύχουν. Και τέλος, να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και το ΖΙΚΑ, το συζητήσαμε και στη ψήφισμα βέβαια, αλλά σας ευχαριστούμε για τη σχετική υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει σχόλια. Nobody from the Commission? Ah, sorry. Αν δεν είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Yeah, good morning. Um... Καλή σας ημέρα. Μάνφρετ ε, Ρόζενστοκ από τη Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντο Environment. Ε, κάποια σχόλια, μια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταθέσει ακόμα πρόταση για την αναθεωρήση του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου. Βλέπουμε και θεωρούμε ότι αυτή η αναθεώρηση αποτελεί μια ευκαιρία να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσει και να εφαρμοστούν οι πολιτικέ προτεραιότητε τι οποίε είχαμε συμφωνήσει για την 7 περίοδο. Προκειμένου να δώσουμε μια όθηση στην ανάκαμψη, στην ε, ανάπτυξη και για να αντιμετωπίσουμε και τι εξωτερικέ προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Στη συζήτηση αναφέρθηκαν κάποιε εξ αυτών. Η πρόταση από πλευρά μα προβλέπεται στα τέλη του τρέχοντο έτου. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Και κοιτώντα και το σχέδιο έκθεση, αναφέρεται διάφορα ζητήματα όπω η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων μέχρι τα μέσα του 2016 και διάφορα ε, σχετικά έργα για μια πρώτη αξιολόγηση, για παράδειγμα, της πρωτοβουλίας αυτής που θα πρέπει να δεδεθεί. Λίγη υπομονή λοιπόν σα ζητώ μέχρι ότου ολοκληρωθεί η πρότασή μα. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο γνωμοδότηση, ασφαλώ σα ευχαριστούμε και από περιβαλλοντική σκοπιά να σα πω ότι είναι σημαντικά τα θέματα τα οποία θίγονται από τον εισηγητή σας ευχαριστούμε και για τα άλλα σημαντικά ζητήματα τα οποία υπογράμμισαν διάφοροι βουλευτές. Ασφαλώς, όλα αυτά θα τα λάβουμε δεόντως υπόψη για την ε, πρότασή μας που θα καταθέσουμε μέσα στο έτος. Μιλήσατε για το θέμα της ενσωμάτωσης της ένταξης των ορίζοντα 2020, το θέμα της μεταρρύθμισης των διαστατικών ταμείων, την αγροτική πολιτική και νομίζω ότι εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι πέρα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως το live, η ενσωμάτωση παραγόντων για το περιβάλλον, για την κυκλική οικονομία, για να αναφερθώ και στο πακέτο που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του προπολογισμού. Και νομίζω ότι εδώ θα βάλω τελεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Καμπούς, για τα τελικά σχόλια στη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους και για το ύφος των, των παρεμβάσεων. Κύριε Γραμματικάκη, πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε και θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και να συνεννοηθούμε. Γιατί δεν νομίζω ότι απέχουμε πολύ στις απόψεις μας. Κύριε Γκέρλινγκ, η συζήτηση για τους ε, γενικούς πόρους που δεν είναι θέμα της Επιτροπής ε, σίγουρα θα πρέπει να είναι τμήμα των ιερών αγελάδων που κανένας δεν μπορεί να αγγίξει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι στο θέμα. Ε, κύριε Τόρβαλ, συμφωνώ ότι οι αγαθές προθέσεις, αν δεν συγκεκριμενοποιηθούν σε έργα, είναι όπλο για το διάβολο. Οπότε θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες ε, να φοδιάσουμε αυτές τις αγαθές προθέσεις με πηξίδα, με αστρολάβο, για να μπορέσουμε να πλέψουμε προς μια σωστή κατεύθυνση. Τις υπόλοιπες απορίες νομίζω ότι τις έλυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά τα σχόλια πάντως ε, να είστε βέβαιοι θα τα λάβω υπόψη στην περαιτέρω επεξεργασία του εγγράφου μου. Σας ευχαριστώ. Μην ξεχνάτε το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι η 5η Απριλίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα γίνει στις 26 Απριλίου, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 15 Ιουνίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έκθεση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες προστατευμένες περιοχές. Όπως θα θυμάστε, οι συντονιστές αποφάσισαν να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανταλλαγή απόψεων με θέμα την έκθεση σε ό,τι αφορά την πρόοδο για τη θέσπιση θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών στα πλαίσια της οδηγίας, της οδηγίας πλαίσιο για τη στρατηγική για τις θάλασσες. I uh, Ακούω ότι η Μαριάν Μπέρνινγκ προϊσταμένη της υπηρεσίας για την ποιότητα της ε, ατμόσφαιρας και των ε, νερών, του νερού, δεν είναι παρούσα. Ε, αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μπορούσε να την καταστήσει ή αν πρέπει να περιμένουμε. Okay. I don't know if we... Ε, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιο να ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμέσω ή αν πρέπει να περιμένουμε. Α, okay. ah, μόλι έφτασε. Πολύ σας ευχαριστούμε. Με συγχωρείτε που σας πιέζω σήμερα. Θα σας περιμένουμε. Οκ, Miss Εντάξει, κυρία Βένινγκ, είμαστε λίγο πιεστικοί σήμερα, γιατί ξεκινήσαμε νωρίτερα, αλλά όταν είστε έτοιμοι θα σας δώσουμε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πραγματικά μας τρέχουν, αλλά ζητώ συγγνώμη για τη δική μου καθυστέρηση, να σας πω καλημέρα και να κάνω κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις ε, σε σχέση με την έκθεση που δημοσιεύτηκε για την πρόοδο που επιτύχαμε για τη θέσπιση προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε η ανθρώπινη ζωή και η ευζωή εξαρτάται και από τη διοπικιλότητα. Η ωκεανή είναι το 90% των οικοσυστημάτων του πλανήτη. που κατοικούνται είτε από είδη θαλάσσια, είτε από πτηνά, είτε από φυτά και υπολογίζεται σε 50-58% του συνόλου της ζωής στην γη και κάτω από την επιφάνεια των ωκεανών. Ωστόσο, οι μελέτε μα δείχνουν ότι οι ωκεανέ και οι ακτέ αντιμετωπίζουν σοβαρέ απειλέ από τι πολλαπλέ πιέσει, του παράγοντε πιέσεων που δέχονται αυτή τη στιγμή. Την υπερεκμετάλλευση των ε, ληφτικών αποθεμάτων, την ρήπανση, την, ε, ε την διάδοση οξέων στου ωκεανού και την καταστροφή συστημάτων. Το 66% των θαλασσίων οικοσυστημάτων ε, στον κόσμο ε, από τα οποία εξαρτάται και η ζωή μας, είτε έχουν υποβαθμιστεί, είτε αντιμετωπίζονται με τρόπο μη βιώσιμο. Η UNESCO υπολογίζει ότι το 2100, εάν δεν προβλέψουμε σημαντικές αλλαγές, πάνω από τα μισά θαλάσσια είδη του κόσμου μπορεί να έχουν εξαφανιστεί. Άρα οι θαλάσσιες περιοχές που θα πρέπει να προστατεύονται, όπως έχουν ονομαστεί στα αγγλικά MPAs, ε, είναι αναγνωρισμένο εργαλείο για να προσπαθήσουμε να αναστρέψουμε αυτήν την ανησυχητική τάση, για να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματά μας και τα θαλάσσια αποθέματα. Τα αποκατεστημένα οικοσυστήματα μπορούν να προσφέρουν τις σοβαρές υπηρεσίες που συνήθως ε, δίνουν, όπως την, ε, τα τρόφιμα, την ψυχολογία, τον τουρισμό, την ε, περιβαλλοντική ανάπτυξη και βεβαίως τα ωφέλη είναι όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και ε, οικονομικά. Το δίκτυο Natura 2000 υπολόγισε τα ωφέλη αυτά σε 1,5 δις ευρώ ετησίως που θα μπορούσαν να προκύψουν μόνο από τα στοιχεία του 2011. Ο αριθμός αυτός όμως θα μπορούσε να διπλασιαστεί. Εάν διπλασιάσουμε και το δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών. Και αν φτάναμε το 10% τότε, πραγματικά θα διπλασιάζονταν, θα διπλασιάζονταν τα οικονομικά ωφέλη. Την 1η Οκτωβρίου πέρσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί για, την, ε, για τον καθορισμό των ε, προστατευόμενων θαλασσίων περιοχών στην Ευρώπη. Το άρθρο 21 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Θαλάσσια Στεργική τα προβλέπει αυτά. Ο στόχος να έχουμε τέτοιες εκθέσεις είναι να υπάρχει μια βασική γραμμή για τους βουλευτές για τις ε, θαλάσσιες περιοχές συγγνώμη, και για τα σχετικά μέτρα, ώστε να έχουμε και στρατηγικά προγράμματα από τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Ήδη τα χρειαζόμαστε φέτος το Μάρτιο, για να μην πω σήμερα, θα πω αύριο. Η έκθεση καταγράφει τον εντοπισμό των θαλάσσιων περιοχών στην Ευρώπη ως το 2012, εξετάζει την οικολογική ε, σύνοχη των ευρωπαϊκών δικτύων των θαλάσσιων αυτών περιοχών και καθορίζει τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη των κατομελών στην ε, ένταση των προσπαθειών τους για να ορίσουν, να διαχειριστούν και να παρακολουθήσουν αλλά και να επιβάλλουν την ισχύ των ε, προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών. Εξήβραμε ότι το 2012 5,9 σχεδόν 6% των θαλασσίων νερών ε, καλύπτονταν, ε, αφορούσαν προς τα επόμενες περιοχές. Τα 2 τρίτα ε, στα πλαίσια του Natura 2000 ήταν τέτοια, τέτοια σημεία και το υπόλοιπο 1 τρίτο ήταν εθνική περιοχές που ορίζονταν από το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Και τα δύο είδη των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, του Natura 2000 ή τα εθνικά, είχαν να κάνουν και με, περιφε... με θαλάσσιες περιοχές σε περιφερειακό επίπεδο. Προστατεύονταν από περιφερειακές συμβάσεις. Υπάρχει λοιπόν κάλυψη στις βόρειες θάλασσες περίπου 80% ενώ η χαμηλότερη κάλυψη ήταν στη Μακρονησία. Ε, υπήρχε μεγαλύτερη κάλυψη παράκτια και στο Πέλαγος ενώ η κάλυψη από, θαλάσσιες, από προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές ε, στην ε, απόσταση πάνω από 12 μίλια από την ακτή είχαμε 40% κάλυψη. Η έκθεση βρίσκεται τα δίκτυα των MPA στην Ευρώπη, δεν είναι οικολογικός συνεκτικά. Παρόλο που κάποιες περιοχές ε, στην Βόρεια Θάλασσα δείχνουν ότι αρχίζουν να συγκλίνουν προς τα σωστά πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη από οικολογικής άποψης, δεν ευσταθούν όσο θα έπρεπε. Εάν αυτό συνέβαινε, θα πολλαπλασιαζόταν ο αντίκτυπος του στην αποκατάσταση των προϋβαλλοντικών θεμάτων. Η Ευρώπη λοιπόν έχει ήδη επιτελέσει σημαντική πρόοδο ορίζοντα αυτέ τι προστατευόμενε θαλάσσιε περιοχέ και σύμφωνα με τι διεθνεί δεσμεύσει που έχει αναλάβει. Όμω πρέπει να συνεχίσει να ε, ε, επεκτείνει το δίκτυο των θαλασσίων περιοχών με περισσότερους οικοτόπους που να καλύπτονται και με την τόνωση των δικτύων των MPA. Τι κάνουμε για να στηρίξουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη στην επιδίωξη των στόχων μας. Πρώτα απ' όλα προωθούμε την πλήρη και ε, διεξοδική εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα γνωρίζετε το MSFT την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, για τα πτηνά και τα οικοσυστήματα επίση. Αυτέ οι οδηγίε προβλέπουν αυστηρά νομικά πλαίσια για τον ορισμό και τη διαχείριση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών. Η ελοποίηση αυτών είναι ζωτική σημασία για να πετύχουμε. Οπότε το να συμπληρώσουμε και να καθορίσουμε το θαλάσσιο μονοπάτι του δικτύου Natura 2000 είναι μια ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ ε, στηριζόμαστε και από την ε, κοινή αλληλευτική πολιτική που συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένε διατάξει για τη διευκόλυνση του ορισμού μέτρων τη αλληλεία, τα οποία είναι αναγκαία για τη διαχείριση των MPA. Το να προβλεφθεί χρηματοδότηση είναι κάτι ακόμη που πρέπει να περάσει από τα κράτη-μέλη, διότι υπάρχει και το πρόγραμμα LIFE, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θαλάσσια ε, Επίση το ΜΑΡΕΣ που χρηματοδοτείται από το ΛΑΕΚ, χρηματοδοτήθηκε από το 2009 στο 2014 και αυτό συνέβαλε σημαντικά στην επέκταση του ισπανικού δικτύου Natura 2000 και των προστατευόμενων περιοχών. Το αποτέλεσμα είναι ότι καλύπτεται το 8% των ισπανικών υδάτων. Επίση, θέλουμε την πρόθεση τη έρευνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα προγράμματα που τρέχουν για να στηρίξουμε την ε, θέσπιση ενό συνεκτικού δικτύου MPA και επίσης χρειαζόμαστε πρόσφατα αποδεικτικά στοιχεία για τα κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη από τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Αναπτύσσουμε μια ευρωπαϊκή συμβέλεια μεθοδολογία για να αποτιμήσουμε την συνέπεια του δικτύου των MPA και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διεθνή φόρα για τις MPA είναι ήδη ε, αρκετά αποτελεσματική όπως συνέβη στον ΟΗΕ πρόσφατα όταν συζητήθηκε η βιωσιμότητα και η προστασία των ε, θαλάσσιων αποθεμάτων σε παράκτιες και τουριστικές περιοχές. Όπως βλέπετε πολλά λοιπόν γίνονται προκειμένου να βελτιώσουμε τα δίκτυα MPA στην Ευρώπη και η διάσκεψη για τους ωκεανούς στη Χιλή το 2015 βρήκε τον Επίτροπο Βέλα να υπόσχεται ότι η κάλυψη 10% ε, θα επιτευχθεί στην Ευρώπη στο 2020 όπως προκύπτει από τη Σύμβαση για την Θελέσσια Επιπικιλότητα και τον βιώσιμο στόχο για το 2025. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιτρέψουμε την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι άκοπες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών ήδη έχουν ε, δώσει κάποια αποτελέσματα. Έχουμε περισσότερα προστατευόμενα μέρη από το 2012, το χρόνο αναφοράς για την εκθεσή μας, ως το τέλος του 2014 λοιπόν. Το θαλάσσιο δίκτυο Natura 2000 κάλυπτε περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ε, κάτι περίπου αντιστοιχεί στο 5% των θαλασσίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με 4% το 2012. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και ε, είμαι εδώ στη διάθεσή σα για τι ερωτήσει σα. Σα ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο, η κυρία Γκέρλινγκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία ερώτηση έχω να κάνω. Νομίζω ότι είναι συνεκτικότητα η έκθεση, την καλωσορίζω και προφανώ είμαι και από ένα κράτο μέλο που περιτριγυρίζεται από υδατά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό για μα και χαίρομαι ιδιαίτερω που σημαίνει το πρόοδο με 17% των υδάτων του Ρημένου Βασίλειου να καλύπτονται πλέον από μια τέτοια MPA. Και έχουμε επίση και χώρια εθνική νομοθεσία που ε, προδιαγράφει την προστασία σε πολλά ιδέα. Μία ερώτηση να κάνω όμως για το μηχανισμό της χρηματοδότησης, κυρίως σε ό,τι αφορά και το e MFF. Υπό πίεση βρίσκεται το τομείο αυτό. Γιατί επηρεάζει και την αλληλεία σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που έχει σε ό,τι αφορά την κοινωνιστική πολιτική. Είχαμε λοιπόν από 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους διάφορες υποχρεώσεις οι οποίες ε, στα είδατα γύρω από το Ενωμένο Βασίλειο παρουσιάζουν δυσκολίε, όσο και αν καλωσορίζουμε τη γενικότερη σύμφωνια, γιατί είναι πολύ μεικτή η αλληλεία. και οι υποχρεώσεις για την εκφόρτωση μας προβληματίζουν. Άρα, μεγάλο τμήμα των προδιαγραφών θα σήμαινε μεγάλες αλλαγές σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης. Και αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσον το EMFF όπως έχει σήμερα και η διαδικασία εκχώρησης η οποία αποφασίστηκε στο προηγούμενο κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες αλίευσης. Κατά πόσον λοιπόν αυτά έχουν νόημα σε ό,τι αφορά τη γενικότερη χρηματοδότηση των MPAs και κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οποιοδήποτε πρόθεση να τα εξετάσει όλα αυτά για να δει κατά πόσον αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο EMFF προδιαγράφονται και έχουν ως σκοπό και εξυπηρετούν τους σκοπούς του MPA και όχι γενικότερα την αλληλεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση έχω να κάνω και από τον τομέα της ε, αλίας της Ολλανδίας. Ξέρουμε τα όσα προδιαγράφουν οι σχετικές προδιαγραφές και την Natura 2002. Στο άρθρο 3 της οδηγίας αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων και θα πρέπει να εξετάσουν την αποδοτικότητα σε ό,τι αφορά τα μέτρα αυτά. Στη σχετική οδηγία, στο Natura 2000 και στο Habitat, ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι αποδοτικά τα μέτρα αυτά. Είναι μεγάλα τα ποσά που δαπανώνται. Θα θέλαμε να μην κάνουμε λοιπόν τα ίδια λάθη και σε αυτή την οδηγία σε ό,τι αφορά την περίοδο 2012 και 2020 σε ό,τι αφορά την Βόρειο Θάλασσα περιορίζονται οι ελευτικέ ικανότητες και δυνατότητες της ε, Ολλανδίας. Ποια είναι λοιπόν η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της αλίας και μήπως αυτό α, ε, περιορίζει τις δυνατότητες των θαλάσσιων περιοχών και σε ό,τι αφορά τις ε, περιοχές Natura 2000 στην Βόρειο Θάλασσα Είδα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλες περιορισμούς οι Και τι γίνεται με τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές όπου έχουν ανακάμψει τα αποθέματα των κομπαδιών. Τι θα γίνει σε αυτές τις περιοχές. Θα εξετάσει και εναλλακτικέ ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεθόδους αλίευσης για παράδειγμα οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και που σέβονται την βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Κυρία Έγκστρομ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενημέρωση. Έχω μερικές ερωτήσεις. Καταρχήν, αλία στις ε, προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες. Συνήθως ε, οι ελληνικές δραστηριότητες ε, με μηχανότρατες ή πολύ επιθετικά ελιαυτικά εργαλεία λαμβάνουν χώρα σε πολλές περιοχές του Natura 2000. Στη Δανία, για παράδειγμα, αυτό ισχύει για τα μύδια ή για τα οστρακόδερμα ε, στην Γαλλία. Πώς λοιπόν τόσο επιζήμιες αλληλευτικές δραστηριότητες επιτρέπονται σε προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες όταν όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αντιβαίνουν στην οικολογική προστασία αυτών των περιοχών. Και τώρα πιο μακροπρόθεσμα για τις ε, θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες. Ο στόχος υποτίθεται ότι θα έχει υλοποιηθεί το 2010 αλλά αναβλήθηκε τελικά για το 2020 για πολιτικούς λόγους η υλοποίηση του στόχου για το ποσοστό το επιθυμητό των MPAs. Η ε, επιστημονική κοινότητα όμως διεθνώς ζήτησε κάλυψη 30% από τέτοιες θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες, παγκοσμίω μάλιστα, και όχι μόνο 20%. Ε, είναι απαραίτητο για τη διατήρηση και την αποκατάσταση του, του θαλάσσιου κεφαλαίου είναι σημαντικό για την ε, σταθερότητα και την βιωσιμότητα. Ποιος είναι ο στόχος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το ποσοστό κάλυψης στον ορίζοντα 2030 και πώς θα συμβιβαστεί αυτό με την ανάπτυξη παράλληλων τομέων που στηρίζουμε θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ποσοστό κάλυψης που να εξασφαλίζει τη συντήρηση των αλληλευτικών ειδών που θέλουμε να προστατεύσουμε. Για παράδειγμα, ναυτικές ζώνες προστατευόμενες με απαγόρευση οποιοδήποτε δραστηριοτήτων εξόριξης. Ε, έτσι θα προστατεύσουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα και θα εξασφαλίσουμε και εκτός των συνόρων τους κάποια οικονομικά ωφέλη. Βέβαια, οι προστατευόμενε θαλάσσιες ζώνες ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτω από το 0,5% του συνόλου των θαλάσσιων προστατευόμενων ζωνών. Ενώ η Αυστραλία έχει 30% κάλυψη τέτοιων ειδικών ε, προστατευόμενων ζωνών. Πώς θα εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη τέτοιων θαλάσσιων προστατευόμενων ζωνών και ιδιαίτερα των ειδικών ε, πάρκων προστατευόμενων ώστε να αναχαιτήσουμε την απόλυτη επικοινότητας. Ευχαριστώ κύριε Σαφρόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή για την ενημέρωση. Θα κάνω ερωτάσεις, ερωτήσεις που ίσως να έχουν ήδη καλυφθεί, κάποιες γενικές ερωτήσεις και μετά μια συγκεκριμένη παρατήρηση. Ε, οι γενικές ερωτήσεις είναι πώς η Ευρωπαϊκή Τροπή σκοπεύει να προχωρήσει σε επίπεδο ε, νόμιμων δράσεων των κατομελών μελών που επί χρόνια δεν έχουν ε, καλύψει κάποιες από τις αδυνομίες τους το δίκτυο των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών όπως ε, υποδεικνύει η Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των θαλάσσιων πάρκων στα χαρτιά, χαρτιά με πάρκα από τα οποία έχουν οριστεί σε συμφωνίε και σε ε, ε πράξει, αλλά δεν έχουν καμία πρακτική εφαρμογή. Έπρεπε να προστατεύονται κάποιες θαλάσσιε περιοχέ, όμω δεν υπάρχει τελικά στην πράξη καμία πραγματική προστασία αυτών. Η Επιτροπή το επενήχθη μόλι. Μπορεί να μα πει ποια μεθοδολογία θα χρησιμοποιηθεί για μέτρα που, προστατεύονται, που προτείνονται για τις προστατευόμενες θαλάσσιε περιοχέ ώστε να βελτιωθεί και η οικολογική του συμβολή και να μπορέσει να βελτιωθεί συνολικά το ποιοτικό επίπεδο των θαλάσσιων ε, νερών της Ευρώπης. Το άρθρο για την κοινή ελευθερική πολιτική προβλέπει τη θέσπιση θαλάσσιων περιοχών βάσει τη οικολογική του ε, σκοπιμότητα. Ε, βάσει του άρθρου 8 λοιπόν τη Συμφωνία για την Κοινή Ελευθερική Πολιτική έχει προβλεφθεί κάτι ανάλογο. Και τα ποσοστά κάλυψης και όλους ιδιαιτέρως η Μεσόγειος. Στη Μεσόγειο το αριθμητικό στοιχείο της έκθεσης 9,7% κάλυψη μας φαίνεται σωστό, διότι 9,7% είναι πολύ κοντά στο στόχο του 10%. Γνωρίζουμε όμως ότι εντός του αριθμού αυτού υπάρχει και το επέλαγος μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας 750.000 περίπου χιλιόμετρα, το οποίο 7.500 ε, χιλιόμετρα που δεν έχει κανένα είδος προστασίας. Εδώ λοιπόν δεν ε, υπάρχει καμία νομοθετική πρόβλεψη για αυτό το μεγαλύτερο καταφύγιο, το λεγόμενο πέλαγος, ε, δεν υπάρχει κανένα είδου πρόβλεψη. Είναι μια από τι ευρύτερε περιοχέ στη Μεσόγειο που θα έπρεπε να καλύπτονται. Το δεδομένο του 10% λοιπόν, που είναι το σύνολο του τι συμβαίνει στα νερά τη Ευρώπη, να το θεωρούμε ω συνολική κάλυψη, γιατί υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ θαλασσών στην Αδριατική έχουμε 2%, στο Ιόνιο 1,6%, στο Αιγαίο 2,6%. Η εξισορρόπηση γίνεται προφανώς από άλλες θάλασσες όπου υπάρχει καλύτερη κάλυψη. Όμως η κατάσταση παραμένει δραματική σε θάλασσες όπου υπάρχει υπεραλίευση ή υπάρχει μεγάλος αντίκτυπος από την πανεπιστήμια παρουσία ή από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπου η υπαρχει μεγαλος αντικτυπος απο την ανθρωπινη παρουσια η απο ανθρωπογενεις δραστηριοτητες οπου η κάλυψη το τεράστιο περιοχών είναι χαμηλότερη. Ελπίζω λοιπόν να δούμε στο ένα ελάχιστο όριο κάλυψη. Μήπω μπορεί να προκληθεί αυτό στο επίπεδο των επιμέρου λεκανών, ώστε να μπορέσουμε ακόμη και σε μια συγκεκριμένη λεκάνη να υπάρχει μια ικανοποιητική κάλυψη έστω 5-6%. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συμφωνήσουμε εκ των υστέρων. Ευχαριστούμε. Κύριε Σπεριάνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα μας είπαν. Με ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εάν ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα μπορούσε να δει τα θέματα αυτά από με την Αλία και η Επιτροπή Περιβάλλοντος η δική μας να τα δει αυτά με την Αλιευτική ε, Επιτροπή ενδεχομένως. Αναφερόμαστε τόσο ή άλλως στην ίδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ και φαίνεται ότι αυτές οι αποφάσεις έχουν στρατηγική σημασία και για τους δύο τομείς, και της Αλίας και του περιβάλλοντος. Είμαι απολύτως για τη χρησιμότητα και το ρόλο των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών για την προστασία και τη συντήρηση των ειδών μας, αλλά ακόμη και για το ρόλο που μπορούν να έχουν στην διαχείριση των ηχθικών, των ελληνικών αποθεμάτων, ιδίω εκεί που υπάρχει έλλειψη ή απειλές. Οι αλληλείς, όπως έδειξαν οι καλές πρακτικές των θαλάσσιων περιοχών που λειτουργούν εύρυθμα, συμμετέχουν και θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες. Αυτή ήταν η πρώτη μου λοιπόν παρατήρηση. Η δεύτερη είναι πέραν των άλλων δύο στην ίδια γραμμή με ω με αυτό που ζήτησε προηγουμένω ο συνάδελφο Αφρόντε. Δύο παρατηρήσεις έχω δηλαδή. Η πρώτη είναι αν το δεδομένο, το αριθμητικό για τι επιφάνειε που καλύπτονται από θαλάσσιε θαλάσσιες περιοχές ε, παρουσιάζει όντως ε, έλλειψη ομοιογένεια. Δηλαδή, ε, περι, θαλάσσιες περιοχές πιο προστατευμένες από άλλες, όπου το ποσοστό των θαλάσσιων περιοχών ε, είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή δεν θα μπορούσαμε να προτείνουμε μια αρχή περιφερειοποίησης όπως υπάρχει στην κοινή ελεκτική πολιτική, διότι είναι λίγο παράλογο να έχουμε περιοχές θαλάσσιες με 2% κάλυψη και άλλες όπου φτάνουμε στο 20%. Εάν οι θαλάσσιες περιοχές είναι όντως περιοχές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ακριβώς και για την αποκατάσταση των ε, αλληλεκτικών, των εχθικών αποθεμάτων, θα ήταν χρήσιμο να λάβουμε υπόψη αυτή την ε, πιθανή αρχή της περιφερειοποίησης. Και η δεύτερη παρατήρηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι για το καταφύγιο Πέλαγος όντως δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή θαλάσσια περιοχή για όλη την Ευρώπη. Είναι μια διακρατική συμφωνία αυτή που το προστατεύει. Όμως, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωρίζει ότι αυτό το εγχείρημα που είναι ε, ιδιαίτερα φιλόδοξο αλλά έχει μείνει στα χαρτιά είναι ακριβώς μόνο μια θεωρητική συμφωνία πραγμα... παρά μια ε, περιοχή που μπορεί να εφαρμοστούν κανόνες. Όχι μόνο για την Αλία αλλά και για όλες τις άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που θα μπορούσαν να πλήξουν κυρίως την προστασία των κοιτοειδών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φαρίας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι πολύ σωστά είπε εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι παράκτιε ζώνε ε, τελούν υπό απειλή. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη και σύντομη ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρούσα κατάσταση στα νότια της Πορτογαλίας, στο Αλγκάρβε, εξαιτίας ε, του τουρισμού και της αλίας. Αυτή τη στιγμή και στη ζώνη του Αλγκάρβε γίνεται πιθανή διερεύνηση για, για πετρέλαιο. Αυτό όμως απειλεί τις ε, ακτές και έχουν υποβληθεί αναφορές και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άμεση πάυση των διερευνητικών εργασιών για την, ε, ε, για την ε, ανέβρεση κοιτασμάτων πετρελαίου. Φαντάζομαι θα γνωρίζει αυτό το αίτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς μπορούμε λοιπόν να προστατεύσουμε από τέτοιες δραστηριότητες ε, την παράκτια ζώνη του Αλγάρβε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κυρία, κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι από την Κροατία και θα ήθελα ολόκληρη η, η Αδριατική να ανακηρυχθεί εθνικός ρημός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θαλάσσιο πάρκο και τι το αξίζει πραγματικά. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε και να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες αυτών που ζουν σε θαλάσσιες περιοχές ή ζουν από τη θάλασσα. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς σκοπεύει να συνδυάσει την προάσπιση και προστασία των θαλάσσιων πόρων, αλλά και την προστασία ταυτόχρονα της αλληλευτικής δραστηριότητας, που είναι από τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε τις συνέπειες της σχετικής νομοθεσίας, αλλά και τη μεταβατική περίοδο που έχει κροατεί για το 2014, κάτι που οδήγησε σε ε, έξοδο από την δραστηριότητα των αλλιέων μικρής κλίμακας. Ε, χιλιάδες άνθρωποι έχασαν την αλλιευτική τους άδεια και έτσι στερήθηκαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν μία ε, μακραίωνη παράδοση που μάλιστα θεωρείται και πολιτιστικό αγαθό στην Κροατία. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε πρωτοβουλία ώστε η ελία μικρής κλίμακα στην Κροατία να ανακηρυχθεί ως πολιτισμικό αγαθό. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν εξετάζει τη δυνατότητα να γίνουν κάποιες νομοθετικές αλλαγές στα πλαίσια της μεταρρυθμίσης και της αλληλευτικής νομοθεσίας, ώστε να ληφθούν υπόψη κάποιες ιδιαιτερότητες και να θεσπιστούν κάποιες εξαιρέσεις στη νομοθεσία για συγκεκριμένες αλληλευτικές δραστηριότητες. Επίσης θα πρέπει αυτή, οποιαδήποτε τέτοια ελευτική δραστηριότητα να έχει τη λιγότερη δυνατή αρνητική συνέπεια για τη θάλασσα, τους θαλάσσιους πόρους και την προστασία των αλευτικών πόρων. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ θερμά όλους για τις ερωτήσεις σας. Τις καταγράψαμε και ελπίζω ότι θα δώσω ικανοποιητικές απαντήσεις. Θα ξεκινήσω με το EMFF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας στα πλαίσια της μικτής διαχείρισης με τα κράτη-μέλη για το χαρακτηρισμό και τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων ζωνών. Πρόκειται για κονδύλια και για ένα ταμείο στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κρατημέλη και γίνεται επιμερισμό στα επιχειρησιακά προγράμματα. Τα επιχειρησιακά προγράμματα τα συζητάμε με τα κρατημέλη και επισημαίνουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά εναπόκειται στα κρατημέλη σε τελική ανάλυση να λάβουν τις αποφάσεις για το κατά πόσο θέλουν να, τα περιλάβουν, να τις περιλάβουν ή όχι. Εδώ πάντως ε, έχουμε πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε Γι' αυτό και έχουμε συνεχείς επαφές με τα κράτη-μέλη και συζητούμε το πώς κατά τη γνώμη μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια ώστε να εξυπηρετήσουμε και να προστατεύσουμε το περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα και άλλα οικονομικά συμφέροντα όπου δει. Τώρα έρχομαι σε ένα ζήτημα που επανειλημμένως αναφέρθηκε από τους ευρωβουλευτές το κατά πόσο δηλαδή οι προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες σχετίζονται με τη διαχείριση της αλίας και την κοινή αλληλευτική πολιτική. Όπως ξέρετε, στα πλαίσια της κοινής αλληλευτικής πολιτικής υπάρχει το άρθρο 11. Αυτό το άρθρο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν χωρίς να περιορίζουν ε, πλήρως ε, τις οικονομικές και ελευτικές δραστηριότητες. Γνωρίζουμε ότι για πολλά κράτη-μέλη το θέμα της αλλίας με μηχανότρατα, για παράδειγμα, ε, προβληματίζει και τα κράτη-μέλη θα πρέπει είτε να, έχουν, να εφαρμόζουν τέτοιες δραστηριότητες με μηχανότρατα είτε με τρόπο που θα είναι συμβατό με το στόχο των θαλάσσιων ζωνών προστασίας ή να απαγορεύσουν ακόμη και κάποιες τέτοιες δραστηριότητες. Αλλά να πω και επαναλαμβάνω στα κράτη-μέλη να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν υπόψη όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και μία θαλάσσια προστατευόμενη ζώνη δεν είναι αποκλειστική ζώνη μίας χώρας. Συνήθως καλύπτει χωρικά τα πολλών χωρών. Οπότε θα πρέπει να γίνει και συντονισμός μεταξύ των χωρών που έχουν κοινή τέτοια θαλάσσια προστατευόμενη ζώνη. Και τα μέτρα στη συνέχεια υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξετάζονται στις αρμόδιες επιτροπές για να εξεταστεί κατά πόσο θα ε, εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο ή όχι. Συνήθως ε, εφαρμόζουμε τη συνοπτική διαδικασία, την fast track όπως λέμε, που είναι και πιο γρήγορη, παρόλο που μερικές φορές είναι πιο χρονοβόρα από ό,τι ακούγεται, γιατί είναι πολλές οι που θέλουν τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη πριν συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα. Πάντως υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν το άρθρο 11 της κοινή ελευτικής πολιτικής. Ένα συναφές ζήτημα αφορά τη συμφιλίωση των στόχων της περιβαλλοντικής προστασίας και της αποκατάστασης και διαχείρισης αυτών των ζωνών με την γαλάζια ανάπτυξη που είναι επίσης στόχος μας. Η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ είναι ιδιαίτερα προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο της γαλάζιας ανάπτυξης, αλλά θεωρούμε ότι δεν αλληλοαποκλείονται οι δύο στόχοι της αποκατάστασης και διαχείρισης των ζωρών και της γαλάζιας ανάπτυξης. Απλώς ε, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες και να εφοδιαστούμε με τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τους δύο στόχους. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι ε, της ε, θαλάσσιας χωροταξίας που υιοθετήσαμε πέρυσι. Εκεί όλες οι δραστηριότητες ε, που λαμβάνουν χώρα σε θαλάσσιες ζώνες, ακόμη και σε προστατευόμενες τέτοιες θαλάσσιες ζώνες, θα πρέπει να είναι συντονισμένες σε κρατικό επίπεδο, ώστε οι συνέπειες μέτρων για, τη, για, τα, για τα τα εμπορικά ή για την ενέργεια ή για τον τουρισμό να λαμβάνονται υπόψη και να ευθυγραμμίζονται με το στόχο των ε, θαλάσσιων προστατευόμενων ζωνών. Οπότε η οδηγία πλαίσιο για τη στρατηγική της θάλασσας είναι επίσης ε, ένα εργαλείο που έχουμε για να εξακριβώσουμε την υλοποίηση των θαλάσσιων μας στόχων ώστε να έχουμε ένα καλό επίπεδο προστασίας και στα παρακτή μέχρι το 2020, αλλά και σωστή και επαρκή κάλυψη για τις θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες. Σε ό,τι αφορά τώρα τους πιο μακροπρόθεσμους στόχους. Επί του παρόντος είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με την επίτευξη προόδου. Αυτή μάλιστα η πρόοδος επιταχύνεται ή έχει επιταχυνθεί την τελευταία διετία. Και έχουμε, θα έχουμε το στόχο κάλυψης 10% μέχρι το 2020 για τις θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες. Και πριν ε, περάσουμε στους μακροπρόθεσμους στόχους, να μην ξεχνούμε αυτό το χρονικό ορίζοντα και ταυτόχρονα μην ξεχνούμε ότι μέχρι το 2020 πρέπει να υλοποιήσουμε ποσοστό κάλυψης 10%. Κάτι που προϋποθέτει μεγάλες προσπάθειες από τα κράτη-μέλη. Όπως είπα, έχουμε τακτικό διάλογο με τα κράτη-μέλη και έχουμε τα βιογραφικά σεμινάρια. Ένα από αυτά αφιερώνεται στις θαλάσσιες ζώνες. Και εκεί εξετάζουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να επιταχύνουμε το χαρακτηρισμό και πρώτα απ' όλα τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων ζωνών. Γιατί δεν μιλούμε μόνο για θέσπιση, χαρακτηρισμό μια ζώνη ω θαλάσσια προστατευόμενη ζώνη, αλλά το θέμα είναι να γίνεται και σωστή η οικολογική διαχείριση αυτή τη ε, θαλάσσια προστατευόμενη ζώνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να το εφαρμόσουν. Γιατί αν δεν έχουμε μια οικολογική συνοχή, τότε δεν θα δρέψουμε τους καρπούς των θαλάσσιων προστατευόμενων ζωνών και για την υλοποίηση αυτών των στόχων σχεδιάστηκαν, οπότε θα ήταν κρίμα να το στερηθούμε. Ε, αυτό το έργο είναι πολύ δύσκολο και σίγουρα δεν είναι ακόμη κάτι κεκτημένο. Θα πρέπει να αντιληφθούμε τι σημαίνει το κριτήριο της οικολογικής συνοχής. Πάντως συνεχίζουμε τις προσπάθειες από κοινού και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος προκειμένου να εκπονήσουμε μεθοδολογίες για να αντιληφθούμε καλύτερα τα κριτήρια της οικολογικής συνοχής και να τα εφαρμόσουμε. Επίσης έχουμε θέματα όπως ε, αντιπροσωπευτικότητα, επάρκεια, ε, διασυνδεσιμότητα. Όλα αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να εφαρμοστούν και εμπράκτος και να γίνουν και λειτουργικά. Επίσης, και αυτό ίσως να καλύπτει και κάποιες από τις ερωτήσεις για την κάλυψη και το αν είναι επαρκής. Είπα στο τέλος της παρουσίασής μου ότι κοιτάζουμε την βιοποικιλότητα πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας. Αυτό ξέρετε ότι στα πλαίσια της διαδικασίας του ΟΗΕ βρίσκεται σε εξέλιξη με, προσ... με προπαρασκευαστικές συζητήσεις που θα δουν την υλοποίηση μιας συμφωνίας βάσει του UN CLOS για την προστασία των θαλάσσιων περιοχών που ξεπερνούν, που ξεπερνούν τα εθνικά όρια, την εθνική δικαιοδοσία. Βέβαια είναι μια διαδικασία που μπορεί να είναι και μακροσκελέστερη, πιστεύω όμως ότι στο τέλος θα καθορίσει την μακροπρόθεσμη θεώρησή μας για αυτό το θέμα με μια ενιολογική κιόλας ε, ε, πανοπλία που ετοιμάζεται. Νομίζω ότι άκουσα μια ερώτηση για την έρευνα και τις ανάγκες της. Ναι, Ήδη στα πλαίσια του Horizon 2020 υπάρχουν κονδύλια για την έρευνα. Μάλιστα χθε το βράδυ πήγα σε μια παρουσίαση κάποιων από των ερευνητικών ιδρυμάτων για να γίνει επιλογή και είναι σαφές ότι πραγματικά, όπως ξέρουμε, Ξέρουμε λίγα πράγματα για τους ωκεανούς στην πραγματικότητα. Περισσότερα ξέρουμε για τη σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης παρά για τους ωκεανούς κάποιες φορές. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε ένθερμα να στηρίξουμε αυτή την ε, άποψη με τα ε, προβλεπόμενα κονδύλια αλλά και τα μελλοντικά βάση του Horizon 2020. Θα μπορούμε να συμβάλλουμε πολύ. Όχι μόνο ε, από την άποψη των χρημάτων που διαθέτουμε στην Επιτροπή αλλά και τις συνεισφορές των κρατών μελών. Το πιο σημαντικό είναι αυτά να χρησιμοποιούνται με τρόπο συνεπή. Αν όλοι πηγαίνουν και κάνουν αυτό που θέλει θα, και, λένε, και ανακοινώνουν απλώ εγώ θα κάνω το ένα και ο άλλο το άλλο, δεν μα βοηθούν. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι οι διαφορετικέ ερευνητικέ προσπάθειε να συνδυαστούν και να βεβαιωθούν ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Τέθηκε ένα θέμα για την νομική δράση. Έχετε δίκιο. Πρέπει να το δούμε για τον καθορισμό των προδευόμενων ε, θαλάσσιων περιοχών. Πρέπει να, το, να ανελάβουμε κάποια σχετική δράση. Ήδη κάποια πιλωτικά προγράμματα τρέχουν και περιμένουμε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα από κάποια κάτι μέλη. Υπάρχει όμως και το δεύτερο batch, όπως το ονομάζουμε, η δεύτερη φουρνιά, με έναν μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών που και αυτό θα παρακολουθήσουμε πώς προχωρεί. Για την ε, Μεσόγειο τέθηκαν συγκεκριμένε ερωτήσει. Το ποσοστό συνολικά είναι υψηλό στην κάλυψη, αλλά αν δει κανεί επιμέρους περιοχές, η συνολική κάλυψη των περιοχών είναι πολύ χαμηλή. Αυτό είναι κάτι που μας αφορά και εμάς και πρέπει να το κοιτάξουμε βάσει της σύμβασης της Βαρκελόνης συζητήσεις ε, και συνεργασία υπάρχει με τις τοπικές αλληλευτικές οργανώσεις και τις περιφερειακές αλληλευτικές ενώσεις για να βεβαιωθούμε όχι απλώς ότι θα αυξήσουμε και θα βελτιώσουμε την ε, διαχείριση των αποστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, αλλά ότι θα βεβαιωθούμε ότι και η πίεση των αλληλευτικών μέτρων περιορίζεται για κάποιες περιοχές που μπορεί να κινδυνεύουν. Έχετε δίκιο. Η κάλυψη εκτός των ειδικών περιοχών βελτιώνεται. Και δεν συζητούμε πλέον μόνο μεταξύ ε, των διάφορων οργανισμών των περιφερειακών και τοπικών, αλλά των μερών της σύμβασης της Βαρκελόνης, τα κατημέλη, το δίκτυο Κοκονέτ. που ασχολείται με τον καθαρισμό των δικτύων στη Μεσόγειο. Και υπάρχουν κάποια μέτρα που ε, ήδη προβλέπονται, αλλά τα κάτι μελη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Η συμμετοχή της DG Mare, της Γενικής Διευθυνσής Mare, ξέρετε τις απόψεις του τρόπου μας, Οπότε θα συνεχιστεί η προσπάθεια. Ήδη έκανα την, τον συσχετισμό μεταξύ του Ταμείου για την Αλία και τη Θάλασσα και του άρθρου 11. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι δύο στόχοι να οδεύσουν σε σύγκληση για την ε, Έχουμε τις μελέτες αντεκτύπου εργαλεία. Έχουμε τον ειδικό σχεδιασμό και άλλα όργανα στη διάθεσή μας. Πρέπει να τα αξιοποιήσουμε αυτά πρώτα πριν προβλέψουμε καινούργια. Ελπίζω να κάλυψα τα πάντα. Ελπίζω να κάλυψα λοιπόν όλη την ξηρά, αλλά μάλλον δεν έχω καλύψει. Και να εκείνη στη διάθεσή σας για τις ερωτές απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ε, πρωινή συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε σήμερα το απόγευμα στις 3. Σας ευχαριστώ. Only with the coordinators at 3 o'clock and Στις συντονιστές. Ε. Members of committee. Thank you. Στις 3 και μετά συνεχίζουμε στις 4. Ευχαριστώ πολύ και καλό διάλειμμα.